Euh, euh, Παίρνω το λόγο γιατί είμαι ο εισηγητής για ε, τα θέματα, τα συναφή θέματα εμπορίου στην Επιτροπή ΙΝΤΕ ε, και θα ετοιμάσουμε την ε, έκθεσή μας μέσω του Προέδρου Ιντα είχαμε ρωτήσει, είχα ρωτήσει λοιπόν ακριβώς α, αυτά τα πράγματα την νομική υπηρεσία και τώρα παίρνουμε την απάντηση διότι θεωρούσα ότι από νομική άποψη ε, θα ήταν, ότι θα ήταν παράξενο τέλο πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει αν θέλετε Εμπορικέ σχέσεις με αυτή την περιοχή να έχει διαφορετική θέση από τους άλλους εμπορικούς εταίρους. Ε, κοιτάξτε, όταν έγινε η συμφωνία ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Μαρόκου, ο κύριος Ζελίκ που είναι τώρα διευθυντή της ε, ε, Παγκόσμιας Τράπεζας, είχε πει ότι αυτή ε, έπρεπε να αποκλειστεί η Δυτική Σαχάρα βάσει των κανόνων του Ηνωμένου, των Ηνωμένων Εθνών τέλος πάντων θα μου πείτε άλλα τα εμπορικά θέματα, άλλα τα πολιτικά θέματα αλλά προφανώς δεν μπορούσαμε να δώσουμε εμπορική απάντηση αν δεν είχαμε τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας ή την πολιτική αν δεν είχαμε υιοθετήσει πολιτική θέση σχετικά με το τι θέλει ο κόσμος της Δυτικής Σαχάρας. Τώρα υπάρχει μια επιχείρηση που λέγεται Αζούρα, γαλλικά κεφάλαια που εξάγει πάνω από 100.000 τόνους ντομάτες του Μαρόκου, από το Μαρόκο. Αλλά ένα μέρος αυτών των 100.000 τόνων ντομάτας προέρχεται από τη Δυτική Σαχάρα. Προς το παρόν λοιπόν δεν έχουμε βέβαια στοιχεία αριθμητικά για το τι προέρχεται από τη Δυτική Σαχάρα για να δούμε ποια είναι η σχέση με το, την ποσότητα που προέρχεται από το Μαρόκο και δεν ξέρουμε αν κερδίζει αν θέλετε ή τι κερδίζει από την εμπορική αυτή συναλλαγή ο λαός της Δυτικής Σαχάρα. Σαχάρας δεν ε, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προσδιορίσουμε το, το χώρο παραγωγής και πώς πρέπει να το λάβουμε υπόψη ή όχι. Για μένα λοιπόν υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. η οχι για μενα λοιπον υπαρχουν πολλα ερωτηματικα και δεν μπορούμε να πάρουμε θέση για τη συμφωνία Μαρόκου Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν ξέρουμε, έχουμε απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Και χαίρομαι που το ίδιο υποστηρίζει και η νομική υπηρεσία. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει εμά, αν θέλετε, σε πολιτικό επίπεδο επίπεδο είναι ποιο είναι το πολιτικό συμφέρον των ο, ανθρώπων που ζουν στη Δυτική Σαχάρα. Να υπενθυμίσω μόνο νομικές φύσεις ερωτήσεις, αν δεν υπάρχουν άλλες να δώσω το λόγο στον κύριο Πάσος και κατόπιν θα ανοίξουν και τις πόρτες. Κανείς θα θέλει το λόγο, λέω. Για τις απαντήσεις παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για να... Για να απαντήσω το πρώτο ερώτημα του κυρίου Λάιενς. Αν η απάντηση είναι όχι στο πρώτο ερώτημα, τότε τι θα συμβεί. Λοιπόν, εγώ είπα η πρώτη ερώτηση πρέπει να είναι η υφιστάμενη συμφωνία σύνδεσης που ισχύει εδώ και 10 χρόνια εμφαρμόζεται, ισχύει και για τη Δυτική Σαχάρα ή στα εφαρμόζεται για τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας. Μετά από 10 χρόνια η Κομισιόν θα πρέπει να μας πει αν καλύπτει η Δυτική Σαχάρα και τα προϊόντα Αν που ναι, τότε το δεύτερο ερώτημα έχει νόημα. Γιατί τότε θα ρωτήσουμε σε ποιο βαθμό τα συμφέροντα και οι επιθυμίες του λαού της Δυτικής Σαχάρας λαμβάνονται υπόψη από το Μαρόκο. Αν μας πούν όχι, η τωρινή συμφωνία σύνθεσης δεν ισχύει για τη Δυτική Σαχάρα, τότε δεν μπορούμε να θέσουμε δεύτερο ερώτημα. Τώρα για αυτά που είπε ο κύριος Μποβέ, τον ευχαριστώ που αναφέρθηκε στην επιστολή Ζελίκ του 2004. Εκεί οι Ηνωμένε Πολιτείε πράγματι στην επιστολή αυτή απέκλεισαν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ε, με την Αμερική βέβαια ε, Μαρόκο Αμερικής ε, Ηνωμένων Πολιτειών απέκλεισαν την εφαρμογή της λοιπόν στα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας τώρα από εκεί και πέρα όντως το Μαρόκο θα πρέπει να δώσει απαντήσεις και όχι η Κομισιόν. Ωραία, αυτό είναι γεγονός. Εγώ, σε εμάς όμως θα απαντήσει η Κομισιόν η οποία γνωρίζει και την ε, συμφωνία σύνδεσης που ε, εφαρμόζεται. Αλλά το, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε εμείς άμεσα ή να έρθουμε εμείς άμεσα επαφή με το Μαρόκο. Δεν είναι δικός μας συνομιλητής του Μαρόκο. Ωραία, σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις αυτές. Κύριε Κουράσοπο της Νομικής Υπηρεσίας, ε, παρακαλώ, ας ανοίξουμε τις πόρτες τώρα, να μπουν όλοι και ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Τη δημόσια συζήτηση πλέον. Ο πρώτος ε, που θα πάρει το λόγο θα είναι ο κύριος Φοντάνα, αλλά ας περιμένουμε ένα λεπτό για να μπουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.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 Possiamo riprendere? Bene, allora. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Κατόμη τη συζήτηση που είχαμε με την ε, νομική υπηρεσία, η Επιτροπή και οι αρχέ του Μαρόκου ολοκλήρωσαν ε, τις διαπραγματεύσεις το Δεκέμβριο του 2009. Βάσει τη συνθήκη λειτουργίας λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύναψη τέτοιου είδου ε, συμφωνία υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η συμφωνία καθορίζει μια πιο ευρία απελευθέρωση των αμοιβών ανταλλαγών γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων. Έτσι λοιπόν η γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα έδινα καταρχήν το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Φοντάνα και κατόπιν θα ακούσουμε και του εκπροσώπου, τον, κύριο, μάλλον τη Κομισιόν, τον κύριο Κλάρκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. στο έργο που υλοποιούμε, κυρίως ε, στις συζητήσεις με διάφορα μέλη και της Επιτροπής Γεωργίας, συνάντησα ε, μια ιδιαίτερη ανησυχία, κυρίως από μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις νότιες χώρες της Ευρώπης για αυτή τη συμφωνία με το Μαρόκο. Καταρχήν θα έχουμε άμεση απελευθέρωση του 45% των εξαγωγών και θα φτάσει το 70% σε 10 χρόνια και 55% των εισαγωγών. Μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό μέρος αυτών των εισαγωγών παρουσιάστηκε ως τμήμα των προκυπευτικών. ακριβώς ό,τι αφορά αυτές τις εισαγωγές ή ανησυχίες τόσο μελών του Κοινοβουλίου, κυρίως Ισπανών, Γάλλων, Ιταλών, οφείλεται στο γεγονό ότι αυτές οι εισαγωγές θα ήταν ανταγωνιστικές, σημαντικά ανταγωνιστικές, ε, έναντι των δικών μας προϊόντων. Κυρίως αναφέραμε σε συγκεκριμένα προϊόντα. Και τέτοιου είδους συμφωνίες ακούσαμε μεταξύ άλλων ότι τίθεται και το νομικό ζήτημα για τη Δυτική Σαχάρα. Δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε περαιτέρω ερωτήσεις, ακόμη και αν φαίνεται να αποκλείεται η Δυτική Σαχάρα, θέλουμε να έχουμε κάτι οριστικό, μια οριστική τοποθέτηση, γιατί εμείς ε, δεν θεωρούμε ε, ότι είναι το ίδιο έτσι λοιπόν, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε πράγματι να δημιουργήσει προβλήματα στους δικούς μας παραγωγούς, γιατί όπως είναι προφανές, ο ανταγωνισμός που γίνεται από μια χώρα που έχει παραμετρούς ποιότητας διαφορετικές και φυσικά κατώτερες σε σχέση με τις δικές μας ε, και αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και μικρότερο κόστος παραγωγής θα δημιουργούσε προβλήματα στους δικούς μας ευρωπαίους παραγωγούς. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε και το θέμα του εργατικού δυναμικού που εργάζεται στο Μαρόκο και είναι διαφορετική κατάσταση εκεί σε σχέση με το τι επικρατεί στην Ευρώπη και μιλάμε και για μείωση του κόστους ε, και της βαριάς παραγωγής. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το περιβαλλοντικό θέμα και το θέμα της διατροφικής ασφάλειας, γιατί από τη σκοπιά της ε, υγείας και της υγείας των φυτών υπάρχουν ε, κατάφορες αποκλήσεις σε σχέση με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ορισμένων ε, ειδών παρασιτοκτόνων που ίσως απαγορεύονται στη δική μας επικράτη ενώ αντίθετα επιτρέπονται στο Μαρόκο. Υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά τον έλεγχο των ροών και την ορθή εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων εισαγωγή. Και πρέπει να, έχουμε, να λαμβούμε υπόψη και αυτό το παράγοντα, δεν πρέπει να τον απαξιώσουμε, ούτε να τον υποτιμήσουμε. Πρέπει να λάβουμε και ε, υπόψη και τους δασμούς ε, ε, στις τιμές εισαγωγής. Πολλές φορές... Ε, Έχουμε επίσης προσπάθειες ε, απάτης και παρουσιάζονται ορισμένα προϊόντα να έρχονται από κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται κάποια τρίγωνα, χρησιμοποιούνται κάποια τρίγωνα και έχει ε, χρησιμοποιηθεί αυτός ο τρόπος ε, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των ποσοστώσεων. Έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι δεν ε, λαμβάνονται υπόψη επαρκής ε, οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ε, για το εργασιακό και μάλιστα όταν μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχουμε τόσο σοβαρή οικονομική κρίση. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι τη στιγμή που η γνωμοδότηση δεν θα λάβει υποστήριξη η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που είναι επί της ουσίας ε, αρμόδια επιτροπή ακούσαμε και τον συνάδελφο Μποβέ ε, δεν θα λάβει καμία γνωμοδότηση από την Επιτροπή Γεωργίας. Ε, αυτό για να σας παρουσιάσω και πώς έχει διαδικασία. Και να πω ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο Μποβέ, γιατί επισημάνθηκε το ζήτημα των ε, Ηνωμένων Πολιτειών ε, το 2004 οι Ηνωμένε Πολιτείε είχαν ε, αποκλείσει τη συμμετοχή της Δυτικής Σαχάρας και μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό περισσότερο για την Αλία αλλά έχει δίκο βάρος και για τη Γεωργία. Αυτά τα εδάφη έχουν δικό βάρος. Έτσι λοιπόν Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω αυτή την πρώτη συζήτηση ενώ στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική αλλά και λεπτή γιατί μιλάμε για μια συμφωνία που θα μπορούσε να είναι σημαντική για το μέλλον της δικής μας οικονομίας, κυρίως από γεωργική σκοπιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Λορέντσο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η γνωμοδότηση. Να σας υπενθυμίσω ότι το σχέδιο της γνωμοδότησης θα παρουσιαστεί στις 14 Μαρτίου και στη συνέχεια θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 28 Μαρτίου. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ελίζα Πετιάγγελ καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους προλαλήσαντες. Όλα αυτά που ήδη ελέγχθησαν θα ήθελα να τα τονίσω, υπογραμμίσω και εγώ. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι η Κομισιόν έχει ε, προετοιμάζει μια ολόκληρη σειρά τέτοιου είδους διμερών συμφωνιών που σίγουρα θα επηρεάσουν τα νότια κράτη-μέλη της Ευρώπης. Πρόκειται και για ντομάτες αλλά και για πολλά άλλα προϊόντα που παράγονται ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν πολύ να προσέξουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια τέτοιου είδους εμπορικού εμπορικών ε, στα πλαίσια τέτοιου είδου εμπορικών συμφωνιών και για να τα αποφασίσουμε αυτά και να κρατήσουμε μια κάποια ισορροπία είναι, θα πρέπει πρώτα πρώτα να ε, έχουμε κάποιους στόχους ένα στόχος είναι να υποστηρίξουμε τις φτωχότερους λαούς του πλανήτη από την άλλη μεριά είναι να υποστηρίξουμε και την γεωργία την ευρωπαϊκή ε, θα ήθελα επίσης να ήξερα ε, κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια κάποια μελέτη ή μια, μια μελέτη αντικτύπων τρόπων την για τις συμφωνίες αυτές. Δηλαδή και για τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δει πώς επηρεάζονται τα προϊόντα. Βεβαίω ορισμένα πράγματα μπορεί θεωρητικά να ακούγονται σωστά, αλλά υπάρχουν και πρακτικά κάποιες δυσκολίες. υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα στις, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας θα ελέγχονται αυτά τα standards. Ε, τι θα γίνει με το περιβάλλον αν υπάρχουν κατάλοιπα από τα φυτοϊγειονομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τα λοιπάσματα κτλ. Τι θα γίνει με αυτά. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες πώς αξιολογούνται μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας. Ε, εμείς φαντάζομαι ότι εδώ στην Επιτροπή μας θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα και να καταλήξουμε σε μια ενιαία θέση και ο κύριος Μποβέ καλά κάνει και τονίζει ορισμένα πράγματα. Βεβαίω δεν έχουμε και πολλές δυνατότητες. Ε, ε, ε, θα πούμε ναι ή όχι δηλαδή στο τέλος, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι αν είναι δυνατόν να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα, να θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων και να σκεφτούμε πώς επιτυχάνουμε τους στόχους μας βεβαίως χρειαζόμαστε εμπόριο βεβαίως χρειάζεται προστασία Ευρωπαϊκή Γεωργία συγχρόνως βεβαίως πρέπει να βοηθηθούν οι φτωχοί λαοί που ζουν δίπλα μας ε, και υπάρχουν και κάποιες τεχνικές πτυχές τύπου standards πρότυπα κτλ τα οποία πρέπει και αυτά να δούμε ευχαριστώ πολύ Herbert Dorfman Πρόεδρε, για την ε, διάσταση εξωτερικής πολιτικής του θέματος αυτού ήδη τα είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσον ε, και πώς μπορούμε να διαπραγματευόμαστε με μία χώρα που δεν είναι μέλος της Αφρικανικής Ένωσης και μεταξύ των Αφρικανικών χωρών ε, έχει και μία πολύ παράξενη θέση λόγω της συμπεριφοράς στην Δυτική Σαχάρα. Τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας δεν ξέρουμε αν συμπεριλαμβάνονται εδώ και βεβαίως αν δεν συμπεριλαμβάνονται τι μήνυμα, τι σινιάλο δίνουμε στις υπόλοιπες αφρικανικές χώρες. Τέλος πάντων, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι βεβαίως υπάρχει και το θέμα των προτύπων και επανειλημμένα το είπε αυτό η Επιτροπή Γεωργίας στο παρελθόν και σε σχέση με άλλα θέματα. Πρέπει να διατηρούνται τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχω και άλλου είδους ανησυχίες. Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν διαπραγματευόμαστε σωστά. Εδώ τι κάνουμε με αυτή τη συμφωνία. Ανοίγουμε την αγορά μας 100% στην ντομάτα του Μαρόκου για προϊόντα τα οποία οποία θα είχαμε εμείς πρόσβαση στην αγορά, δηλαδή, τι να σας πω, αχλάδια μήλα, ξαφνικά μπαίνουν ποσοστώσεις και δει ποσοστώσεις που είναι πολύ πιο χαμηλές από αυτές που θα μπορούσαμε να εξάγουμε εμείς. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Νομίζω ότι ναι, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο διεθνές εμπόριο, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε και οι δικές μας γεωργικές εκμεταλλεύσεις να μπορούν να διαπραγματεύονται τα προϊόντα τους σε άλλες αγορές. Θα πρέπει να είναι ισότιμη η διαπραγμάτευση. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε πλήρως <coughs> τη δική μας αγορά για τα προϊόντα της χώρας με την οποία διαπραγματευόμαστε και να οι δικές της αγορές να μένουν εν μέρη κλειστές για τα δικά μας τα προϊόντα. Δεν είναι καλό το μήνυμα αυτό για, και για τις άλλες συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε με χώρες πιο σημαντικές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ντρεπόμαστε να πούμε ότι υποστηρίζουμε τους αγρότες μας και ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να ανοίξουμε πλήρως τις αγορές μας εάν και οι αγορές των άλλων δεν ανοίξουν πλήρως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χέρμπερτ. Ε, δεν μπορούμε να πληρώσει η Γεωργία τα πλέον εκτήματα που θα επιτευχθούν σε άλλα εδάφη από αυτές τις συμφωνίες. Μάρτιν και μετά και Βοβέ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα κάνω ανάλυση της ε, ε, Προτίμηση μου. Το είπε και ο ίδιο ο πρόεδρο, Δεν πρέπει να τα πληρώσει η Γεωργία οποιαδήποτε παραχώρηση γίνεται στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών και εδώ δεν πρέπει να μιλάμε για αντισταθμίσει. Πρέπει να περασπίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων παραγωγών εδώ. Όταν μιλάμε για μια νέα συμφωνία, εγώ θέλω να αναφερόμαι και στην ισχύουσα και στην ισχύουσα συμφωνία με το Μαρόκο διαπιστώνουμε με σαφήνεια και το λέει ε, και η Όλαφ ότι δεν σέβονται τις ποσοστώσεις και ότι δεν σεβούνται τις τιμές αναφοράς. Έτσι λοιπόν υπάρχει ε, μια αίτηση της Επιτροπής Αναφορών και νομίζω και μια επιστολή με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου που ζητείται από την Κομισιόν να προβεί σε μεταρρύθμιση του κανονισμού του 2007 σε σχέση με τις τιμές αναφοράς και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να τροποποιηθεί αυτή Τόσο ο κανονισμός, καθώς προκύπτει σαφής απάτη και αν δεν είναι αυτοργοποίηση δεν θα δεχτούμε μία άλλη συμφωνία που να ωφελεί περισσότερο το Μαρόκο. Επίσης, ε, θέλουμε να αναφερθούμε στις ε, ξαφείς απαιτήσει ε, που υπάρχουν, στις διαφορές απαιτήσεων που υπάρχουν για τα φυτογειονομικά, τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ισχύει σε τρεις χώρες. Δηλαδή, μπορούν να έρθουν ελεύθερα από το Μαρόκο προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα ίδια παραστοκτόνα τα οποία εμείς επαγαρεύουμε. Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Και εγώ θα ήθελα να προτείνω αυτά να λαμβάνονται υπόψη στην έκθεση και αναφέρομαι στο ότι το Μαρόκο έχει θέσει σε εφαρμογή το πράσινο σχέδιο, όπως το αποκαλεί, για να αυξήσει τα επόμενα δέκα χρόνια την γεωργική του παραγωγή. Μιλάμε για 700.000 εκτάρια που θα τεθούν στην παραγωγή και αυτό θα έχει συνέπειες απαράδεκτες κατά την άποψή μου. Και νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε με κανέναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό τον ανταγωνισμό και πρέπει αυτό να το έχουμε ήδη υπόψη, γιατί αυτό το σχέδιο, το πράσινο σχέδιο όπως το αποκαλούν, ήδη λειτουργεί, μιλάμε για ένα μέλλον 10 ετών και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη, γιατί στο μέλλον πραγματικά θα το δούμε ε, να έχει σημαντικές συνέπειες. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μποβέ, παρακαλώ. Δεν θα ήθελα να επαναλάβουμε εδώ πέρα τη συζήτηση όσον αφορά τα νομικά ζητήματα, τα καλύψαμε πριν από λίγο. Όντως ήμουν εισηγητής για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Για μένα λοιπόν το ζήτημα αυτό το γεωργικό θα πρέπει να το εξετάσουμε από την αρχή του. Δηλαδή, Μιλάμε για διάφορα προβλήματα. Το πρώτο όμω πρόβλημα είναι οι εισαγωγέ, ο όγκο των εισαγωγών. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η συμφωνία αυτή εφόσον να εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε αύξηση 22% εισαγωγές ντομάτας, 150% για τα κολοκύθια, 140% για τα μανταρίνια, για τα αγκούρια και μια τεράστια αύξηση εισαγωγές των φραουλών. 3.500% αύξηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έχει τεράστια δυσμενή επίπτωση για τον αγροτικό πληθυσμό της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καταρχάς την πραγματικότητα αυτή. Τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία σας παρέθεσα είναι οι άμεσες εισαγωγές εφόσον η συμφωνία υπογραφεί αύριο. Μέσα σε τέσσερα χρόνια οι όγκοι αυτοί βέβαια θα παρουσιάσουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής σημαίνει ότι λέμε σε όλους τους γεωργούς στη Νότια Ευρώπη τελείωσε το παιχνίδι, δεν έχετε μέλλον. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το ζήτημα των τιμών και το ζήτημα του σεβασμού των τελωνιακών δασμών. Μπορούμε για παράδειγμα να φανταστούμε ότι έχουμε την αγορά του Περπινιών όπου περνάνε όλα αυτά τα προϊόντα, η επιτήρηση εκεί πέρα δεν γίνεται σωστά. Επομένως μιλάμε για ένα πραγματικό πρόβλημα dumping που υπάρχει όσον αφορά τους φόρους που δεν καταβάλλονται και τις τιμές που καθορίζονται. Όσον αφορά τα φυτο και τα σχετικά πρότυπα, το αναφέραμε η έλεγχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται με τρόπο συστηματικό, δεν είναι αρκετά δυναμική, υπάρχει επομένως σε ένα πρόβλημα. Τέταρτον, υπάρχουν πάρα πολλά εδάφη που δίνονται σε διάφορα επενδυτικά ταμεία όπου γίνονται οι επενδύσεις αυτές οι οποίες οδηγούν στις εξαγωγές αυτές και καταλαβαίνετε ότι οι επενδύσεις αυτές δεν δεν σέβονται καθόλου τα συμφέροντα των τοπικών παραγωγών, των μικρών παραγωγών. Ουσιαστικά οι επενδύσεις που γίνονται από μεγάλες βιομηχανίες ε, εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα. Αναφέρθηκε για παράδειγμα στην εταιρεία Αζουρά, η οποία εξάγει πολύ μεγάλες ποσότητες από ντομάτες και οι εξαγωγές αυτές όμως δεν αποφελούν καθόλου τους μαροκινούς γεωργούς. Επίσης, το ζήτημα έπειτα του εργατικού δυναμικού και αυτό είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα καθόδες. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα σε μια κατάσταση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπραγματευτεί χωρίς να μιλήσει ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έτσι τελικά γίνεται τα πράγματα, δεν ακολούθησε τους κανόνες εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόβλημα αυτό το έχουμε και με το Μερκοσούρ και με τον Καναδά. Κάθε φορά βέβαια για διαφορετικούς τομείς παραγωγής μπορούμε εμεί να συνεχίσουμε να δεχόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απλώ θα περιμένει να μαθαίνει, να ενημερώνεται για τι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής που λαμβάνονται χωρί τη δική του συμβουλή. Γιατί πώ θα καταφέρουμε να μεταρρυθμίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική προ όφελο των γεωργών και των καταναλωτών και των Ευρωπαίων πολιτών όταν έχουμε παράλληλα συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών οι οποίε καταρρύπτουν κάθε προσπάθεια που εμεί, ω ευρωβουλευτέ, έχουμε κάνει για την κοινή γεωργική πολιτική. Γι' αυτό το λόγο στα πλαίσια της ε, έκθεσης που θα κάνω για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, θα προτείνω να καταρρίψουμε να μην δεχθούμε την ε, έκθεση αυτή, τη συμφωνία αυτή και να θέσουμε νέους κανόνες για το μέλλον. Τζορτζ Λέιον και ο κύριος Δανέλης στη συνέχεια. Παρακαλώ, George. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια θα ήθελα να υποβάλω και δεν θα με ακρηγορήσω γιατί κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτά που θέλω να πω κι εγώ. Σε συνδυασμό με την ε, συνεδρίαση που είχαμε και κλεισμένο των θυρών και σε σχέση με αυτά που ζητά αυτή η Επιτροπή από την Κομισιόν, το αν συμπεριλαμβάνεται η Δυτική Σαχάρα στη Συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό να το προσδιορίσουμε αυτό. Πρέπει να κατανοήσουμε αν ε, τα συμφέροντα των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας έχουν ληφθεί υπόψη και Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε σαφήνεια για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα και εγώ ανησυχώ ότι, γιατί δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου και πάλι εδώ ε, ακούσαμε ότι και όπως έγινε με την Μερκοσούρ δεν είχε ενημερωθεί το Κοινοβούλιο, δεν είχε ενημερωθεί για τις συζητήσεις και μας είπαν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη μελέτη αντικτύπου, οπότε καταλαβαίνω ε, δεν μας, ε, λένε ότι ούτε καν μπορεί να γίνει. Συγγνώμη, εγώ δεν το δέχομαι αυτό, γιατί μπορεί κάποιος ε, να καταρτήσει διάφορα σενάρια ε, και να αναλύσει τον αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα. Πρέπει να λάβουμε κάποια απόφαση και πρέπει να καταλάβουμε τι διακυβεύεται εδώ ε, και τι δράση θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω και δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν υπάρχει επίσημη μελέτη αντικτύπου. Έτσι λοιπόν, ε, νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή ως θέμα αρχής να επιμείνει θα έπρεπε και να ζητήσει από την Κομισιό να προβεί σε εκπόνηση αυτής της μελέτης αντικτύπου για να μπορέσουμε να κρίνουμε λογικά αυτά τα θέματα. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η Επιτροπή να αποφασίσει από κοινού με την Κομισιόν για το πώς ε, θα προχωρήσουμε στη σχέση που θα συνάψουμε με την Κομισιόν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ε, μία μελέτη αντικτύπου για να ξυλογήσουμε γιατί αυτό δεν συμφέρει την Ευρώπη ε, γιατί ε, θα πρέπει να υποστηρίζουμε εδώ τη σύναψη συμφωνιών με κάθε τίμημα. Εγώ νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε πρέπει να κάνουμε όσα προτάθηκαν από την νομική υπηρεσία και δεύτερον θα πρέπει να επανέλθουμε στην Κομισιόν και να επιμείνουμε να μας ε, παρουσιάζουν μια μελέτη αντικτύπου προκειμένου να καταλήξουμε και σε κάποιες αποφάσεις. Ο κύριος Δανέλης. Μαρτινός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ένα δύσκολο και ευαίσθητο θέμα που γίνεται πιο δύσκολο για μας αφού δεν μπορούμε να κάνουμε καμία τροποποίηση στις ε, διατάξεις της συμφωνίας. Ε, βέβαια, στα νομικά ζητήματα και στο ό,τι αφορά την Δυτική Σαχάρα δεν θα αναφερθώ. Περιμένουμε όμως κάποιες απαντήσεις από την Κομισιόν. Και συμφωνώ απόλυτα με την ευκαιρία να αναφέρω ότι ε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν και να αποδεχόμαστε τη στάση της Κομισιόν σε όλα αυτά τα ζητήματα τα τόσο ευαίσθητα για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων ε, γεωργών και κτηνοτρόφων, η στάση της σε σχέση με κορυφαία θέματα όπως η Μερκοσούρ, όπως ο Καναδάς ε, και τώρα το Μαρόκο ε, είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε ως ακολουθητές των όποιων ζητημάτων η Κομισιόν θεωρεί ότι προέχουν. Δεν αμφισβητώ ότι πολιτικά είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Και βεβαίως αποδέχομαι ότι μία συμφωνία κρίνεται ε, από το σύνολό της και όχι από, τις, τα επιμέρους. Όσον αφορά όμως τους Ευρωπαίους καλλιεργητές, κυρίως των ε, ε, οποροκυπευτικών, τα συμφέροντα φύγονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό το λόγο και η, στάση μας είναι πολύ δύσκολη. νομίζω ότι και με ευκαιρία αυτήν τη συμφωνία ότι δεν θα πάψουμε να βλέπουμε αμυντικά κάθε φορά όποιο αντίστοιχο θέμα έρχεται αν δεν βρούμε απάντηση, αν δεν βρούμε λύση στην πραγματική στήριξη των πολιτικών ποιότητας και ασφάλειας των αγροδιατροφικών προϊόντων. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων παραγωγών και έτσι θα στηρίξουμε και το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Ε, δεν ξέρω ποια θα είναι η πολιτικά σωστή απόφασή μας. Ε, γι' αυτό το λόγο διατυπώνω σκέψεις και προβληματισμούς περιμένοντας και τις κρίσιμες απαντήσεις από πλευράς Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάρτιν Όσλινγκ. Äh, ναι, υπάρχουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με αυτές τις συμφωνίες και αναφέρθηκαν μερικά. Βεβαίως ζούμε και μια κατάσταση τεράστιων ανατροπών στον αραβικό κόσμο αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό ε, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας, δεν ξέρω. Ορισμένα πράγματα ίσως θα μπορούσαν να αλεχθούν πριν από μερικού μήνες. Δεν μπορούν να αλεχθούν τώρα ή θα πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες για να τα συζητήσουμε στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, ε, η βάση της... Ε, ε, υφιστάμενες συμφωνίες έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, ότι κάποιες εισαγωγές δεν γίνονται βάσει των κοινωνικών, δεν μιλάω για τα στάνταρ ποιότητας, των κοινωνικών στάνταρ που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη από άποψη ε, εργασιακών συνθήκων. Ε, ε, οπότε... Ε, πρέπει να προωθούμε τέ, τέτοιου είδους συμφωνίες και να γινόμαστε συνένοχοι σε τέτοιου είδου κινήσεις. Ίσως ε, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί γιατί υπάρχουν όπως ελέγχθη και πολλές άλλες συμφωνίες που προετοιμάζει η Κομισιόν. Ελεύθερες συναλλαγές δεν λέω ότι δεν μας συμφέρουν, δεν συμφέρουν την Ευρώπη, δεν συμφέρουν τη Γερμανία. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γαρσία Ευχαριστώ, και κατόπιν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι Πιστεύω ότι είμαστε ικανοί όλοι οι συνάδελφοι που πήραμε αυτή τη στιγμή να συμφωνήσουμε στο εξή ότι μιλάμε για μια συμφωνία η οποία θίγει κάποιους πολύ ευαίσθητους τομείς για την δική μας γεωργική παραγωγή. Μιλάμε και για μεγάλες χώρες. Όμως, ε, εγώ πιστεύω ότι για να συμφωνήσουμε στο θέμα αυτό θα πρέπει να εκπονήσουμε το καθήκον μας, ε, να ε, είμαστε υπεύθυνοι. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν με τη συμφωνία αυτή και ορισμένοι συνάδελφοι το έθεσαν πριν πάρω εγώ το λόγο. Το ε, σημερινή. Η σημερινή συμφωνία που ισχύει από το 2003, που επικαιροποιήθηκε με τις διευρύνσεις το 2004 και 2007, ήδη καθόριζε την απελευθέρωση συγκεκριμένων προϊόντων και την ε, βελτίωση της πρόσβασης άλλων ε, μέσω συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και μείωση των τιμών και με την ε, αλλαγή των ποσοστώσεων. Μιλάμε για τη συμφωνία που υπεγράφει το 2003. Ίσως αυτό το πρωτόκολλο δεν ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να υπογραφεί. Ίσως εκείνη τη στιγμή, κατά την έγκρισή του, να έγινε κάποιο λάθος και είδαμε ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν. Όμως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοί να διαβάσουμε το περιεχόμενο της νέας πρότασης και να δούμε πώς τίθενται σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ρήτρα διασφάλισης, όπως είναι η στήριξη σε και από την άλλη, κατανοώ πλήρω και υποστηρίζω την ανησυχία ε, ορισμένων παραγωγών ε, όπως της ντομάτας, παραδείγματος χάρη, ε, για που θα μπορούσε να θίξει ιδιαίτερα αυτό το τομέα η εν λόγω συμφωνία. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να ε, γίνουν οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν και αναφέρομαι και στους έλεγχους για τις ποσοστώσεις και στους έλεγχους για τις τιμές ε, εισόδου. Αν δεν πληρούνται ε, αυτοί οι έλεγχοι, τότε θα πρέπει εμείς να αναλάβουμε δράση για να υλοποιούνται οι έλεγχοι αυτοί. Γιατί είπαν ε, κάποιοι ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την Συμφωνία, αλλά αν δεν υλοποιούνται οι έλεγχοι, ας αναλάβουμε εμεί δράση για να πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, οι τιμέ εισόδου κτλ. Γιατί έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πιο ευαίσθητου ε, τομεί ε, στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνίας. Και Μιλάμε για μια συμφωνία η οποία εντάσσεται στη διαδικασία της Βαρκελόνης και μιλάμε για την προώθηση της ζώνης ελεύθερων συναλλαγών. Έτσι λοιπόν εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να δούμε τα ζητήματα αυτά πιο καθολικά και πιο γενικά. Επιμένω εκ νέου, αναγνωρίζοντας πάντοτε το ότι είναι ευαίσθητα ορισμένα προϊόντα και φυσικά κατανοώντας και την ανησυχία που έχουν ε, ορισμένη παραγωγή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιμείνουμε και να εργαστούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν και να ολοκληρώσουν αυτά τα συστήματα ελέγχων. Και υποστηρίζω, σε είπα κ. Μάτου, για την τροποποίηση του κανονισμού που έχει να κάνει με τις τιμές εισόδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαστάνκο και κατόπιν κύριος Νταντά. Ε, στηρίζω την προσέγγιση ε, του κυρίου Φοντάνα και είμαι πάρα πολύ ευτυχής που την έκθεση επί της ουσίας την έχει ο κύριος Μποβέ στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δηλώνω ρητά κύριε Μποβέ ότι θα στηρίξω ε, τη δική σας προσέγγιση πάνω σε αυτό το πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ε, αναδείχθηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για τα προϊόντα του Ευρωπαϊκού Νότου. Ε, εγώ αν συγκρατώ κάτι από τη λειτουργία μας σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου, είναι ότι ε, αναδεικνύουμε κοινού τόπους ανεξαρτήτως γεωγραφικής προέλευσής μας από τον Νότο, από το Βορρά, από το Κέντρο, από την Ανατολή ή από τη Δύση. Ε, χρησιμοποιήθηκε, μάλλον η φράση κλειδί σε αυτή τη συμφωνία είναι τα αμοιβαία μέτρα ε, ελευθέρωσης. Αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης σημαίνει αμοιβαιότητα, αλλά αμοιβαιότητα όχι ως ρητορικό σχήμα, αμοιβαιότητα είναι της πράγμαση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Το βλέπουμε και σε άλλες περιπτώσεις των εξωτερικών σχέσεων, των εξωτερικών διαστάσεων της αγροτικής πολιτικής. Αναφέρθηκαν πολύ σωστά ε, η, ανάγκη αναφέρθηκε για ισοδύναμες προδιαγραφές, φυτογειονομικές, κοινωνικές, πολύ σωστά είπε ο κύριος Χόισλινγκ, ε, ζητείται το greening της ευρωπαϊκής ε, γεωργίας, αλλά από την άλλη δεν διασφαλίζεται στους κάθε φορά ε, εταίρους μας. Και καταλήγοντας θα ήθελα να πω ότι, κοιτάξτε, η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας του γενικού συμφέροντος, του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος, εν προκειμένου του ευρωπαϊκού γεωργικού συμφέροντος. λοιπόν πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, που ο αρμόδιος Επίτροπος Διεθνού Εμπορίου συμπεριφέρεται με θεσμοπολιτική υπεροψία έναντι του δημοκρατικά νομιμοποιημένου σώματος που λέγεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ευχαριστώ κύριε Μποβέ που συγκατανεύετε σε αυτό που λέω. Πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε αυτόν τον Επίτροπο ότι δεν μπορεί να αγνοεί, να παραβιάζει ο ίδιος με τη στάση του, με τη συμπεριφορά του, με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το ότι είναι θεματοφύλακας του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος. Και αυτό το μήνυμα κύριε Πρόεδρε πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα δηλώνω ότι δεν θα συμφωνήσω στην Ολομέλεια, συμφωνήσω στη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι ε, αυτής της συμφωνίας. Και νομίζω ότι πρέπει να συστρατευτούμε όλοι πάνω σε ένα όχι, προκειμένου να στείλουμε το μήνυμα του δικού μας θεσμικού και πολιτικού βάρους. Είναι θέμα αρχής για την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ σαφή τόσο μας είπατε ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Σε συνέχεια των όσων είπε ο σας, με την ευκαιρία της συζήτησης αυτής της έκθεσης νομίζω θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τη μέθοδο καταρχάς. Γιατί πρόκειται για μια πρώτη από έναν κύκλο συζητήσεων που κάνουμε αυτή τη στιγμή για τις διμερείς σχέσεις και ξέρουμε ότι ακολουθούν και άλλες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις οποίες θα κληθούμε να συζητήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι ως Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν αγώνα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και εκτός Κοινοβουλίου. Στο στερικό του Κοινοβουλίου Ήδη έχουμε χάσει μετά την, ομο, την ομόφωνη ψηφοφορία που είχαμε στην Επιτροπή Γεωργίας και έπειτα στην Ολομέλεια μετά την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ίντα για διάφορα ζητήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση θεσμικής φύσης ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα και καταρχάς να δούμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε περισσότερο με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ίντα, οι οποίοι δεν φαίνεται να συντοποιούν τη διάσταση των ζητημάτων όπως εμείς. Επίσης, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ότι η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν λαμβάνεται υπόψη από έναν επίτροπο, ο οποίος αγνοεί ουσιαστικά το πώς ψηφίσαμε στην Ολομέλεια και επιπλέον μας ρίχνει στην μία ή την άλλη συζήτηση και πολλές φορές θεωρεί ότι είμαστε αδαείς εμείς για κάποια ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι θα πρέπει η δική μας Επιτροπή να θέσει τη στάση μας κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε τουλάχιστον η πολιτική μας τοποθέτηση να γίνεται γνωστή στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το Κοινοβούλιο όμως από την άλλη έχει και μια αρμοδιότητα ελέγχου. Θεωρώ λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να κάνει κάποιες αποστολές Επιτήρηση ελέγχου, για να δει επιτόπου για το πώς εφαρμόζονται και υλοποιούνται όλες αυτές τις συμφωνίες τις οποίες εγκρίνουμε. Πολύ ωραία, ευχαριστώ Μισελ. Ο Thank you, Chair, and Ευχαριστώ πολύ και θα είμαι πολύ σύντομη γιατί ε, έχουν ακουστεί πάρα πολλά από αυτά που ε, θα έλεγα και εγώ και επανελειμμένα ελεγχθεί ότι η Κομισιόν αποφασίζει να κάνει μια εμπορική συμφωνία. Εμείς το μαθαίνουμε εκ των υστέρων και δεν ε, ε, ξέρουμε και πολλά για τη συμφωνία αυτή. Θα μιλήσω και αναφέρομαι εδώ και στις συμφωνίες με το Μερκοσούρ. Εν πάση περιπτώσει ε, είναι πολύ σημαντικό εμείς σαν Επιτροπή Γεωργίας να δηλώ και ως εκπρόσωποι όλων των αγροτών της Ευρώπης να πούμε ότι θέλουμε διμερείς συμφωνίες που ε, όχι μόνο όχι βέβαια να διμερείς συμφωνίες που όπως είπε και ο κύριος Παπαστάμικος να είναι ε, ισορροπημένες και δίκαιες. Ε, προσπαθούμε να πρασινίσουμε τη δική μας γεωργία, δεν κάνουμε το ίδιο και τους εμπορικούς μας εταίρους. Αυτό είναι τουλάχιστον παράξενο. E, Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Το παραδέχομαι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ συχνά έχουν διαφωνήσει με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν ήμασταν υπεύθυνοι για τα θέματα αυτά. Κανεί δεν ζητούσε από εμά να πάρουμε αποφάσει. Ενώ τώρα άλλαξαν τα πράγματα μετά τη θέση σε σχέση τη συνθήκη τη Λισαβόνα και εμεί είμαστε πλέον υπεύθυνοι ενώπιον των Ευρωπαίων αγροτών σε σχέση με τι αποφάσει που λαμβάνονται. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση αυτή Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συμφωνία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους Ευρωπαίους αγρότες. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα αγαθά που θα εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει αυτής της συμφωνία θα ωφελήσουν του καταναλωτές. Βλέπουμε να υπάρχει απειλή σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων αυτών και σε σχέση με τις προϋποθέσεις παραγωγής τους και μάλιστα ποιος παράγει τα προϊόντα αυτά και σε ποιες συνθήκες. Τρίτον, να τονίσουμε ότι τα μεγαλύτερα ωφέλη από τη συμφωνία αυτή θα προκύψουν για τους εμπόρους και για όσους συνάπτουν πολυετής συμβάσεις. Δεν θα υπάρχει όφελος για τους ίδιους τους γεωργούς, ούτε καν για τους ε, γεωργούς στο Μαρόκο, καθώς ε, υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες και ανησυχίες. Και καθώς υπάρχουν τόσες πολλές αμφιβολίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να συμφωνήσει ενώπιον ε, αυτής της συμφωνίας. Κατά την άποψή μου, Όπως σας είπα, επειδή είμαστε συνυπεύθυνοι έναντι των καταναλωτών και των αγροτών για τις ε, αποφάσεις αυτές, ε, θα πρέπει να έχουμε και ανάλογη στάση. Νίκολσον, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, τα σχόλια από τα νότια τμήμα της Ευρώπης. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ακούμε και τους ανθρώπους από τις περιφέρειες που έχουν τις ανησυχίες και συμφωνώ με κάποιες από τις ανησυχίες που ακούστηκαν εδώ. Έχουμε πρόβλημα μέχρι τώρα για το θα πούμε ναι ή όχι με τέτοιες, σε τέτοιες προτάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να διαλέξουμε αυτές που μας αρέσουν και δεν μπορούμε να αυτές που δεν μας αρέσουν. Έτσι λοιπόν συμφωνώ με άλλους που είπαν ότι δεν είναι καλή ιδέα και η Κομισιόν φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα υπέρ των διμερών συμφωνιών που συνάπτουν. Εμείς πρέπει να θέσουμε κάποιες αρχές σε αυτή την Επιτροπή και με βάση αυτές τις αρχές να λαμβάνουμε αποφάσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι κύριοι Φοντανά και Μποβά είναι οι δύο και θα μπορέσουν να, ε, να επιλύσουν το ζήτημα αυτό και φυσικά θα ακολουθήσουμε όσο είπε και ο κύριος Λάιον. Χρειαζόμαστε και μελέτες αντικτύπου. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε στο μέλλον με οτιδήποτε η Κομισιόν μας παρουσιάζει και συμφωνώ και με τον κύριο Κοντανά. Εκτό ε, αν έχουμε κάποιο είδο συνεργασία με την οποία ίντα, ε, τότε δεν ε, θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ορθή οδό, γιατί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των γεωργών. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι ήταν ε, μια ενδιαφέρουσα σειρά ανταλλαγή απόψεων. Να προσθέσω κι εγώ ότι συμφωνώ με όσοι υπόθηκαν του συνέντευξη, να προσθέσω και ένα θέμα μεθοδολογία, ε, τη μεθόδου τη σύναψη διμερών συμφωνιών. Αυτή που θα συνέψουμε σήμερα, ό,τι θα δώσουμε σήμερα στο Μαρόκο, αύριο θα πρέπει να το δώσουμε και στην Ισία και στι υπόλοιπε χώρε. Έτσι λοιπόν η Γεωργία χάνει από τι διμερεί ε, συμφωνίε. Εμεί είμαστε υπέρ των πολυμερών συμφωνιών. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο τώρα στον πρόσωπο τη Κομισιόν, τον κύριο Κλάρκ, για να προσπαθήσει να μα παράσχει όλες ε, τι πληροφορίε που ίσω θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν του βουλευτές. Παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ζητήσω από έναν συνάδελφο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να μας πει μερικά πράγματα για την Δυτική Σαχάρα. Ε, Ε, ε, ε, εμπίπτει το θέμα αυτό στις δικές του αρμοδιότητες και καινούργιες υπηρεσίες που έχουμε. Αλλά τώρα για τα σχόλια που έγιναν από την Επιτροπή σας ξέρω ότι η πλήρη συζήτηση θα γίνει στις 14-15 Φεβρουαρίου όταν θα και τότε θα μπούμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες για τη συμφωνία αυτή όταν θα είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Παρόλα όλα αυτά ας δώσω μερικές πρώτες απαντήσεις σε αυτά που άκουσα. Συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι θα πρέπει το, τη συμφωνία αυτή να τη δούμε στο σύνολό της και όχι ανά και Μόνο έτσι η Επιτροπή σας μπορεί να καταλάβει κατά πόσον ε, πληρούνται τα συμφέροντα των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Γεωργίας αφενός και τα συμφέροντα των φτωχών γειτόνων μας, του Μαρόκου συγκεκριμένα, αφετέρου. Τώρα για το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής. οφείλω να ομολογήσω ότι η συμφωνία αυτή είναι κατά την άποψή μου μετριοπαθής τουλάχιστον όσον αφορά το τι καλύπτει. Θα πρέπει να σημειώσουμε πρώτα πρώτα ότι υπάρχει ήδη μια συμφωνία που ισχύει εδώ και δέκα χρόνια. Αυτή η συμφωνία μέσα στα πλαίσια του πολιτικού πλαισίου των σχέσεων μας με τους μεσογειακούς μας γείτονες ε, προβλέπει αμοιβαία απελευθέρωση γεωργικών προϊόντων. Ο, στις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων ωστόσο δεν ε, είναι ελεύθερο εμπόριο με τις χώρες αυτές. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Και έτσι λίγο λίγο απελευθερώνουμε τις ε, συναλλαγές μας. Ξεκινήσαμε με 30% εισαγωγές από το Μαρόκο τώρα πάμε στο 55% τις εισαγωγές αυτές ε, που δεν είναι λόγο γίνεται πλήρες άνοιγμα των ε, ευρωπαϊκών αγορών από το 30% πάμε στο 55%, 55 για τις εισαγωγές. Τώρα, για το, το συμφέρον του Μαρόκο, Ε, το Μαρόκο άνοιξε 14% των ε, αγορών του σε ευρωπαϊκά ε, συγγνώμη, ε, με αυτή την έννοια εμεί ανοίγουμε στο Μαρόκο 14% των προϊόντων των αγορών μας, 70% ανοίγει το Μαρόκο για μας. Θα πάρει 10 χρόνια αυτό βεβαίως, αλλά είναι Πρόκειται για απελευθέρωση αμοιβαία, ασύμετρη μεν, αλλά που τελικά συμφέρει και είναι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας περισσότερο από ό,τι της του Μαρόκου. Βεβαίως ελέγχθη ότι πρόκειται για ευαίσθητα θέματα, ευαίσθητα προϊόντα όπως η ντομάτα που είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει στη συμφωνία αυτή να αυξήσει την πρόσβασή της την πρόσβαση του Μαροκού κατά 52.000 τόνους ε, σε τέσσερα χρόνια. Και το, άρα το σύνολο της απελευθέρωσης για το Μαρόκο θα είναι 285.000 τόνοι μετριοπαθής αύξηση θα έλεγα της ποσόστοσης για την ντομάτα του Μαρόκου και πολύ βρισκόμαστε ακόμη σε χαμηλότερα επίπεδα ε, από ότι οι πραγματικές εμπορικές συναλλαγές 52.000 ντομάτε, ε, 52.000 τόνοι ντομάτα 8 εκατομμύρια τόνους ντομάτες παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση ετησίως. Απελευθερώνουμε λοιπόν το 0,6% 100, δηλαδή δίνουμε στο Μαρόκο 0,6% της αγοράς μας επιπλέον από ό,τι είχε το Μαρόκο αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν από οικονομική άποψη τι ε, ε, μελέτη αντικτύπου να κάνουμε για το 0,6% της αγοράς. Σίγουρα δεν κλείνει εδώ η συζήτηση, θα γίνουν και άλλες συζητήσεις. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε τη συμφωνία αυτή στη σωστή της προοπτική. Ε, πρέπει να έρθουμε και σε επαφή με τις διάφορες ομάδες, να εξηγήσουμε τα στοιχεία, να τα δούμε με κάποια ψυχραιμία θα έλεγα. Τώρα για άλλα πράγματα για άλλες ανησυχίες που αναφέρθηκαν για τις απαιτήσει του συστήματος ε, γενικευμένων προτιμήσεων um, τα φυτογειονομικά θέματα και τις, ε, ε, τα πρότυπα γιατί ο σεβασμό διαφόρων προτύπων από το Μαρόκο αυτό πρέπει να γίνει και προβλέπονται και κάποιες ε, συμβουλευτικές και διαβουλευτικές δημοκρατικές διαδικασίες αν χρειάζεται κάτι τέτοιο να προσεχθεί περισσότερο επίσης εάν και εφόσον υπάρξει αναταραχή στο εμπόριο που δεν την προβλέπω αυτή τη στιγμή μπορούν να γίνουν επιπλέον συζητήσεις και αναθεωρήσεις Κάποιος τώρα μίλησε και για απάτες και τη διαπτώση παΐστοση απατών από εισαγωγής εξαγωγές. πράγματι το 2007 ο η Όλαφ έκανε σχετικές έρευνες σχετικ... για τα οποροκυπευτικά γιατί υπήρχαν καταγγελίες για απάτες και βρήκαν βρήκε η Όλαφ ένα πολύ χαμηλό βαθμό υπό ε, υποτίμησης αν θέλετε της αξίας των προϊόντων που ήταν γύρω στις 300.000 ευρώ τώρα καταλαβαίνετε ότι 300.000 ευρώ όταν μιλάμε για τέτοιου είδου εμπορικέ, συναλλαγές είναι ασήμαντο ποσό Αυτά είναι τα επιπλέον στοιχεία τα οποία θα ήθελα να αναφέρω εδώ για να δούμε τη συμφωνία αυτή λιγάκι με στο σωστό της πλαίσιο αλλά βεβαίως όπως σας είπα θα γίνουν και άλλες συζητήσεις μαζί σας και ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε υπό το σωστό πρίσμα την οδηγία αυτή. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιάννησεν για να συμπληρώσει ορισμένα πράγματα, ιδιαίτερα σε σχέση με τη Δυτική Σαχάρα. Να, κοιτάξτε, λίγα λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη για το ζήτημα αυτό λοιπόν της Δυτικής Σαχάρας. Μιλάμε εδώ πέρα για τη συμφωνία αυτή, για τα αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα προϊόντα της με το Μαρόκο. Τίθεται λοιπόν και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας και ήδη τίθεται από τη στιγμή που υπάρχει το άρθρο 16 της συμφωνίας που ισχύει ήδη από το 2000, όπου προβλέπεται μία προοδευτική ελευθέρωση των προϊόντων των γεωργικών και των προϊόντων αλίας. Η συμφωνία που συζητάμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίθηκε από, το Ευρωπαϊκό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2009 και είχε ως στόχο να τροποποιηθεί η Συμφωνία Σύνδεσης και ουσιαστικά στόχος το πέρα να τροποποιηθούν κάποια άρθρα και κάποια πρωτόκολλα. Στην Συμφωνία Σύνδεσης γίνεται απλώς αναφορά στο Μαρόκο. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη Δυτική Σαχάρα. Και ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την ε, Συμφωνία με τα μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα. Θεωρείται ότι είναι διοικητική αρχή de facto το Μαρόκο για τη, δίκη, για τη Δυτική Σαχάρα, θεωρείται μη αυτοκυβερνόμενο έδαφος η Δυτική Σαχάρα για τα Ηνωμένα Έθνη. Έτσι λοιπόν σύμφωνα με νομική γνωμοδότηση των Εθνών του Φεβρουαρίου 2002 και με βάση το διεθνές δίκαιο οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τους φυσικούς πόρους, α, τις οποίες συναλαμβάνει μια de facto διοικητική αρχή σε μη αυτοκυβερνόμενο έδαφος, δεν είναι παράνομες δραστηριότητες, αρκεί αυτές να μην αντιτίθεται σε επιθυμίες και τα συμφέροντα του λαού του εδάφους αυτού. Επίσης, η de facto διοικητική α, διοίκηση του Μαρόκο του Μαρόκου προς την Δυτική Σαχάρα καλείται να καλύψει ακριβώς και να σεβαστεί τα συμφέροντα και τις επιθυμίες αυτές. Επομένως, ούτε η αρχική συμφωνία σύνδεσης, ούτε η υποεξέταση συμφωνία προβλέπουν, προβλέπουν συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο, τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Φοντάνα για κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση αυτή. Σημειώνω τις ε, θέσεις που ακούστηκαν εδώ στην Επιτροπή μας ε, και περιμένω και τη συνεργασία όλων για τη σύνταξη της επόμενης γνωμοδότησης, του σχεδίου ε, γνωμοδότησης και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 7 τώρα για να επιτρέψουμε στον συνάδελφο Ταπάτσι ε, να νωρίτερα, η συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Ο κύριος Σταπέτζης λοιπόν είναι ο συντάκτης της νομοδότησης. Αμέσως σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι αυτή η συμφωνία η οποία θα έπρεπε να συναυθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας δεν ε, θα προκαλέσει τόσο έντονες συζητήσεις όπως η συμφωνία με το Μαρόκο. Γιατί δεν πρόκειται για μια νέα συμφωνία. Το 2002 συνήθω μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας προκειμένου να προστατευτούν ε, οι ε, προστατευόμενες ομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δεν έχει ακόμη προετοιμάσει την έκθεσή της, αλλά εμείς προετοιμάσαμε τη δική μας γνωμοδότηση. Στην γνωμοδότηση αυτή προτείνω στην Επιτροπή Γεωργίας να προτείνει, μάλλον να εγκρίνει την πρόταση της Κομισιόν για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας με την Ελβετία για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης. Μόνο δύο σχόλια θέλω να κάνω. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ήδη έχουμε υιοθετήσει την έκθεση του κ. Σκοτέ για την πολιτική ποιότητας και μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας θα υιοθετήσουμε την νομοθεσία για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων. Γι' αυτό προτείνω στην νομοδοτησή μου να καλέσουμε για την υιοθέτηση μάλλον κατόπιν της υιοθέτησης της νομοθεσίας αυτής, η Επιτροπή να αναθεωρήσει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, η Κομισιόν να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να συνάψει τη συμφωνία αυτή με την Ελβετία βάσει της νομοθεσίας. Τώρα, τη δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η βάσεις δεδομένων δεν είναι αρκετά ακριβείς. Αναφέρομαι στι βάσει δεδομένων, ονομασιών προέλευση και γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό σημαίνει ότι το παράρτημα δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή κατάσταση. Οι βάσεις δεδομένων DOR και IBACUS αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του Σεπτεμβρίου του 2009. Γι' αυτό η Επιτροπή Γεωργίας προτείνει στην Κομισιόν να επικαιροποιήσει τα δεδομένα των βάσεων αυτών και να συμπεριλάβει τις νέες ονομασίες προέλευσης και τα νέα προϊόντα που προστατεύονται από γεωγραφική σκοπιά. Προτείνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να δεκτεί η Επιτροπή Γεωργία στην γνωμοδότησή μου με αυτές τις δύο παρατηρήσεις και βάσει αυτών να δεκτείτε τη σύναψη μια νέα συμφωνίας με την Ελβετία. Και μια πληροφορία. Υπήρξαν ε, κάποιες συζητήσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελβετίας, μεταξύ Αυστρίας και Ελβετίας, που ρυθμίστηκαν χάρη στην προηγούμενη συμφωνία για την προστασία, για τις προστατευόμενες ονασίες και αυτές ε, οι διαφορές έχουν ρυθμιστεί. Σήμερα δεν υπάρχει καμία διαφορά, καμία διάνοιξη ό,τι διαφορά της προστατευόμενης ονασίας πρόληψης και της γεωγραφικής ενδείξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Ταμπάτζη. Τώρα, θα ξαναδίνω στο λόγο στον κύριο Κλάρκ, εκτός αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο. Ο κύριος Κλάρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή σαφώς δεν ε, είναι ως ήταν η προηγούμενη συμφωνία που συζητήσαμε. Έχουμε βέβαια και το Μερκοσούρ που ακολουθεί στο μέλλον. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ταμπάτση για την γνωμοδότησή του. Καταγράφουμε όλες τις παρατηρήσεις που κάνει σε αυτή τη γνωμοδότηση και τις οποίες ανέφερε και σήμερα. Η συμφωνία αυτή δεν καλύπτει το αλκοόλ και το κρασί, αυτό καλύπτεται, αυτά καλύπτονται σε εφιστάμενη συμφωνία, η οποία αναθεωρείται σε τακτική βάση, Επομένως, κατά αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι η κάλυψη αλκοόλ και ίνου είναι επικαιροποιημένη. Η συμφωνία αυτή έχει να κάνει με τις ονομασίες προέλευσης, και τις γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν προϊόντα πέραν των, του αλκοόλ και του ίνου. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτικής μας για την ποιότητα και η συμφωνία αυτή προβλέπει ακριβώς αυτή την πλήρη προστασία αυτών των γεωγραφικών ενδείξεων και ελπίζω ότι ε, η Επιτροπή ουσιαστικά θα εγκρίνει την πρόταση αυτή της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Ταπάντζη, όχι. Πολύ ωραία. Τότε μπορούμε να περάσουμε στην προθεσμία κατάσταση τροπολογίων 3 Φεβρουαρίου μεθαύριο. Έτσι λοιπόν κατόπιν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν τη συμφωνία με την Ελβετία. Και τώρα, ας περάσουμε στο σημείο 3 της ημερησίας διάθεσης. Και είναι οργάνωση αγοράς και ειδικών διατάξεων γυρισμένα γεωργικά προϊόντα. Τώρα εδώ θέλω να σας ζητήσω να με προσέξετε. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας με μια παρουσίαση από την Κομισιόν της πρότασης ευθυγράμμισης και απλούστευσης ε, της ΕΝΙΑΣΚΟΑ. Αυτό το εγχείρημα κατέστη απαραίτητο μετά τη θέση ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα που κατέργησε το παλιό σύστημα της Επιτροπολογίας και εισήγαγε ένα άλλο σύστημα με τις λεγόμενες κατεξουσιοδότηση πράξη, δηλαδή άρθρο 290 και τις εκτελεστικές πράξεις του άρθρου 291. Η Κομισιόν παρουσίασε τις κυρίες γραμμές της διαδικασίας ευθυγράμμισης το Δεκέμβριο ήδη όταν συζητήσαμε την ευθυγράμμιση του κοινισμού για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη. Σήμερα η Κομισιόν θα παρουσιάσει την πρόταση ευθυγράμμισης της ενίας ΚΟΑ ε, η οποία είναι πιο πολύπλοκη και ε, Κατόπιν θα δούμε και την πρόταση της χρηματοδότησης της ΚΑΠΗ. Η Επιτροπή προτείνει ε, για την ενία ΚΟΕ. Προτείνει λοιπόν η Κομισιόν για πρώτη φορά τη χρήση του άρθρου 43 παράγραφος 3 της συνθήκης που εισάγει μια διαδικασία όπου μόνο το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις χωρίς καμία εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ λεπτό ζήτημα και από πολιτική σκοπιά και από θεσμική σκοπιά και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και τι ακριβώς συντρέχει από νομική σκοπιά εδώ. Να δώσω όμως το λόγο ε, στον κύριο Ουλκε που θα μας παρουσιάσει τις προτάσεις αυτές. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Ντεκάστρο, είναι πολύ ικανοποίηση. Πολύ μεγάλη ικανοποίηση μου να είναι εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι και σε αυτό το καινούριο κτίριο και φαίνεται ότι έχετε πάρα πολύ καλέ εγκαταστάσει. Ε, σα ζηλεύουμε εμεί στην Κομισιόν για τα κτίρια σα. Αλλά τέλο πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, ήρθα εδώ για να κάνω μια παρουσίαση. Δεν νομίζω όμως ότι πρέπει να μακρηγορήσω, γιατί πολύ μάλλον ε, γνωρίζετε καλά το εγχείρημα αυτό. Είπατε και εσείς ήδη έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις για την ευθυγράμμιση. Εδώ μιλάμε για μια μεγάλη δέσμη μέτρων, ε, ευθυγράμμισης καθώς αφορά την ενιακόα. Έχει πάνω από, περιλαμβάνει πάνω από 300 σελίδες, πάνω από 300 άρθρα, πολλά παραρτήματα. Αλλά για να απλουστεύσω. Περιδημός πρόκειται. Ουσιαστικά εδώ προσπαθούμε να προσαρμόσουμε την εννέα κόστη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, για να προβούμε σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα περνώντας από την παλιά διαδικασία της επιτροπολογίας όπου είχαμε διαχειριστικές επιτροπές και ένα σύστημα ειδικής πλειοψηφίας ε, ε, αν πήγαμε στο Συμβούλιο ή διαφορετικά προβαίνουμε στην εφαρμογή, το σύστημα της κανονιστικής διαδικασίας όπου χρειαζόμαστε ειδική πλειοψηφία υπέρ Όλα αυτά είναι κάτι που πρέπει να τα ξεχάσουμε, να τα αφήσουμε πίσω μα ε, και να περάσουμε στην εποχή τη Λισαβόνα, αν μπορώ να το πω έτσι. Και τώρα για την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να θεωρηθεί επίγουσα. Για τον απλό λόγο ότι έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Απαντά στην ανάγκη σαφήνεια. Η ενιαία ΚΟΑ αν και προσαρμόστηκε προσφάτως το 2007, έχει υποστεί αρκετές τροπήσεις λόγω της μεταρρύθμισης του ίνου το 2008, τις αποφάσεις για τη health check ε, της ΚΑΠ το 2009 και ήδη τώρα βρισκόμαστε σε μια ζούγκλα άρθρων. Αυτό αρέσει πάρα πολύ στους δικηγόρους αλλά όχι στους ε, κοινούς κινητούς. Γιατί δεν είναι βανάγνωστο όλα αυτά. Έτσι λοιπόν το εγχείρημα αυτή τη πρόταση τι είναι, να ενοποιήσουμε ότι έχουμε και να καταστήσουμε επανάγνωστο το κείμενο, να έχει μια δομή που θα επιτρέπει και στου μη νομικού ε, να κατανοήσουν αυτή τη σημαντική νομοθεσία. Νομίζω ότι είναι αυτό σημαντικό να το τονίσουμε. Και επίση, Έχουμε εδώ και ένα στοιχείο διαφάνειας, απλούστευση και διαφάνεια. Αυτή είναι η στόχη αυτού του εγχειρήματο. Κατόπιν. Πρέπει να καταστήσουμε λειτουργική τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και γι' αυτό μπαίνουμε τώρα στο πιο λεπτό τμήμα του εγχειρήματο. Πρέπει να υπογραμμίσω. Στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν επιμένει στο ότι δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με τις αρμοδιότητες. Δηλαδή σε σχέση με τις αρμοδιότητες που έχει σήμερα η Κομισιόν στα πλαίσια της επιτροπολογίας και της διαδικασίας διαχειριστικής επιτροπής, κανονιστικής επιτροπής κτλ. Εδώ δεν ήρθαμε για να αρπάξουμε περισσότερες αρμοδιότητες. Ε, αρέσει η εξουσία στην Κομισιόν, αλλά δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο εδώ. Θέλουμε απλώ να κάνουμε μια προσαρμογή τη νομοθεσίας μας στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και σε αυτή τη διαδικασία έχουμε διατύπωση από τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία δεν είναι τόσο προφανής και αυταπόδεικτη. Εγώ δεν ε, συμμετείχα στις ε, συζητήσεις στο Συμβούλιο, ούτε στις συζητήσεις για τη τακτική συνέλευση, αλλά, αλλά ε, πολλές φορές αναρωτιέται κανείς ε, πώς προκύπτει αυτή η διατύπωση. Κοιτάξτε τώρα, πρέπει να το δεκτούμε και πρέπει να μπούμε σε ένα ιδιαίτερα σχολιστικό εγχείρημα. Κάθε φορά που υπήρχε μια διάταξη με πράξεις κατανάθεση στη Διαχειριστική Επιτροπή ή στην Εγκληστική Επιτροπή, πρέπει να δούμε αν ε, στο μέλλον δηλαδή με τη συνθήκη Αβώνα, θα εμπίπτει στι εκτελεστικέ πράξει ή στι πράξει κατεξιοδότηση. Και στι εκτελεστικέ πράξει ε, που αποκολουθείται η διαδικασία τη διαχειριστική επιστροπή, διαδικασία όπω τη γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε ειδική πλειοψηφία κατά για εμπλοκή. Αυτό είναι γνωστό, το ξέρουν τα κράτη-μέλη. Δεν ε, είναι κάτι καινούριο. Έτσι λοιπόν, ε, με αυτή τη διάταξη, με τις εκτελεστικές πράξεις, έχουμε τη δυνατότητα για την Κομισιόν και μόνο, όπως είναι σήμερα, η Κομισιόν και μόνο, δύναται να λάβει την απόφαση. Δηλαδή εδώ μιλάμε για την εφαρμογή της μείωσης συντολιστών παραδείγματος χάρη στις ποσοστώσεις όταν ε, ξεπερνούν οι αιτήσει στη διαθέσιμη ποσότητα ή για καθορισμό κάποιων εισαγωγικών δεσμών. Ε, Παραδείγματο χάρη, όταν έχουμε τη μέση αναφορά για τα λαχανικά. Αυτά θα πρέπει να τα διαχειρίζεται η Κομισιόν, χωρί επιτροπή. Και περνούμε τώρα στι πράξει κατεξουσιοδότηση. Πράξει εξουσιοδότηση υποτίθεται πως αποτελούν ε, μια τροποποίηση μη ουσιαστική στη βασική πράξη. Όπως αποφασίστηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Για να παρασχεθεί κάποιο πλαίσιο για προσαρμογή αυτών των πράξεων που δεν είναι ουσιαστικές. Ιωνή ε, νομοθετικής φύσεως τις αποκαλούμε και φυσικά αν υπερβαίνει κάτι τέτοιο τότε εμπίπτει στη βασική πράξη. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη σαφή δομή, η κατανομή των εργασιών, βασική πράξη, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεύτερον έχουμε τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση με τα στοιχεία του ελέγχου και της ανάκλησης από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και το τρίτο επίπεδο είναι η διαδικασία της επιτροπολογίας ένα είδος ημι διαχειριστικής επιτροπής. Τώρα, σε αυτό και κάνοντα αυτή τη διάκριση σε σχέση με το τι εμπέπτει στι εκτελεστικέ πράξει και το τι εμπίπτει στι πράξει κατοξιοδότηση, φτάσαμε σε κάτι πολύ δύσκολο, όπω θα το έλεγα. Προσπαθήσαμε με το καλύτερο τρόπο να κάνουμε μία ερμηνεία τι εμπίπτει πού. Και αν ήμασταν ε, πολύ προσεκτικοί, ήμασταν ιδιαίτερα σόφρονες ε, πώ Όποτε είχαμε μία αμφιβολία, προσπαθήσαμε τότε να το θέσουμε σε πράξη κάτω εξουσιοδότηση έναντι της επιλογής άλλη εναλλακτική, δηλαδή εκτελεστική πράξης. Έτσι λοιπόν, προσπαθήσαμε να είμαστε σόφρονες και να διασφαλίσουμε ότι δεν ε, θα παρουσιάσετε εδώ ότι ξεπερνούμε τις διατάξεις της άμονας ε, των άρθρων 290 και 291 για τις πράξεις κατοξιοδότηση. Τώρα, ε, συγγνώμη για τις εκτελεστικές πράξεις, τώρα για τις πράξεις κατοξιοδότηση, όπως ξέρετε έχουμε τη δυνατότητα μόνο η Κομισιόν να πάρει αποφάσεις και οι αποφάσεις αυτές φυσικά μπορούν να, ε, να ε, τύχουν αντίρρησης ε, από το Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο και μπορεί να ε, υπάρχει απόσυρση ή μπορεί να υπάρχει χρονικός περιορισμός της εξουσιοδότησης ή μπορεί να ανενωθεί σιωπηρά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία με την αλλαγή της βασικής πράξης αν αυτό απαιτείται. Έχουμε λοιπόν αρκετά πρακτικά στοιχεία που υπόκειται σε αυτή την ε, κοινή συνεννόηση, έχει τυποποιηθεί συνεννόηση μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιών ε, για να δούμε πώς όλα αυτά θα λειτουργήσουν. Είπα ότι μόνη η Κομισιόν, έτσι το έχει διαρθρώσει η συνθήκη. Δεν ε, είναι βέβαια απαραίτητο ότι αυτό θα ήθελε η Κομισιόν, γιατί αυτό θέτει την Κομισιόν σε μία δύσκολη κατάσταση αν εμείς ε, μόνοι μας, ε, το χάρη, βγούμε στην ανοιχτή θάλασσα και θα αντιμετωπίσουμε μια καταιγίδα η οποία θα έρχεται είτε από ε, τα δεξιά του Συμβούλιο από τα αριστερά από το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό έχει νόημα να διαβουλευόμαστε με εμπειρογνώμονες, με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη και θα διαβουλευόμαστε και με εμπειρογνώμονες από το Κοινοβούλιο. Βέβαια από το Κοινοβούλιο εξαρτάται να αποφασίσει κατά τη δική σας κρίση, δηλαδή πώς εσείς θα εργαστείτε, αυτό θα το αποφασίσετε εσείς. Δεν θα σας δώσουμε καμία συμβουλή, εκτός από το ότι θα προτιμούσα να έχουμε τη γραμματεία από το Κοινοβούλιο ή τους βοηθούς ή όλους τους που ε, θα συνεργάζονται μαζί μας. Τώρα, ο στόχος της διαβούλευσης αυτής ε, είναι προφανής. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ουσιαστικά στοιχεία είναι πάγια. Δηλαδή ότι λαμβάνουμε μία απόφαση που μπορεί να σταθεί σε μία αντικειμενική βάση. Αλλά και κάτι ακόμη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να αποφύγουμε ότι συνεχώς θα προκύπτει μία κατάσταση όπου το Συμβούλιο ή το Κοινοβούλιο θα θεωρείται ότι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά τους όπλα. Δηλαδή είτε αντίθεση είτε την ατομική βόμβα που είναι η ανάκληση της εξουσιοδότησης. Δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και πόσο μάλλον της Κομισιόν να έχει μια τέτοια κατάσταση. Εμείς θέλουμε να έχουμε διαδικασίες που να λειτουργούν μεταξύ Κομισιών, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, έτσι ώστε να έχουμε ε, μία ομελή λειτουργία αυτής ε, της διαδικασίας. Δεν θέλουμε να προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις. Αυτά για τη γενική πρόταση σε ό,τι αφορά την κατανομή των εργασιών μεταξύ εφαρμοστικών διατάξεων, βασικών αξιών, κατεξοδότηση πράξεων κτλ. Και τώρα να έρθω σε ένα θέμα που αγγίξατε κι εσείς, Πρόεδρε, που έχει να κάνει με αυτό το κανθόδες ε, θέμα του 43-3. Δεν ξέρω πού προήλθε. Ούτε εγώ ούτε τη συναδελφή μου συμμετείχαμε σε αυτή τη συζήτηση. Και αν μου επιτρέπετε, εγώ θα προτιμούσα σήμερα να μην υπήρχε. Αλλά υπάρχει. Και επομένως πρέπει ουσιαστικά σε αυτό το σκελετό να δώσουμε και κάποια σάρκα βγήκε από την τουλάπα, πρέπει να ζήσουμε με αυτό και νομίζω ότι ο σκελετός ε, είναι ένα υπόλοιπο του παρελθόντος που είχαμε διαπραγματεύσει κάθε χρόνο, τότε καθορίζαμε τιμές, ποσοστώσεις, έτσι λοιπόν ε, κάπως τυχαία αν θέλετε μπήκε. Τι κάναμε όμως, ε, προσπαθήσαμε να δώσουμε μια ερμηνεία το κύριος τη της Αγώνα για τη συναπόφαση είναι να υπάρξει συναπόφαση για την αγροτική πολιτική και δεν έχει νόημα αν αυτή είναι η κυριαρχή να αφαιρέσουμε ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα και να πούμε «Α, το Κοινοβούλιο τίποτα δεν έχει να πει με τις ποσοστώσει του γάλακτος για τι τιμέ ή για τις ποσοστώσεις τη Ζάχαρη ή για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. οποία έχουν να κάνουν με τη σκόα για το γάλα, για τη ζάχαρη κτλ. Είπαμε λοιπόν, να είμαστε λογικοί. Ας ε, προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια πρόσθετα στοιχεία που να σέβονται το πνεύμα της συνθήκη και του 43.3. Αλλά να μην αγκιστρώνονται πάνω στην ίδια στην πολιτική. Έτσι λοιπόν, αυτό θέλουμε να προτείνουμε στο νομοθέτη, να εφαρμόσει το 43-3 με πολύ μετρημένο τρόπο. Και πρέπει να έχουμε κάποια κριτήρια για την ιδιωτική αποδοματοποίηση του βουτύρου, το χάρη, ε, ή για τη χρήση του αποβουτυρωμένου γάλακτος, ε, για τις ζωοτροφές. Για να το πω ειλικρινά, μη, μιλάμε για μη ουσιαστικά στοιχεία της κοινή αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, εμείς προσπαθήσαμε να το δεκτούμε και προσπαθούμε τώρα εδώ να υποβάλουμε μια πρόταση. Θα έχουμε μια πρόταση που θα παρουσιαστεί για το 43 παραγραφος 3, αλλά προσπαθήσαμε να ζήσουμε εδώ με αυτό το σκελετό που βγήκε από τον τουλάπι. Αυτά νομίζω έπρεπε να πω κύριε Πρόεδρε στο στάδιο αυτό. Θέλουμε να έχουμε μία ταχεία υιοθέτηση της πρότασης αυτής. Γιατί? Γιατί σήμερα όσο λειτουργούμε από την ενία ΚΟΑ, συνεχίζουμε να εμπίπτουμε στην επιτροπολογία τη εφιστάμενη παλιά συνθήκη. Δεν εφαρμόζουμε τη συνθήκη τη Λισαβόνα ε, ω προ την επιτροπολογία, όσο η πρόταση αυτή δεν θα έχει υιοθετηθεί από το συνομοθέτη από τόσου συνομοθέτες, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν σα καλούμε να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατόν στην υιοθέτηση. Να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία για το πακέτο της ποιότητας, το πακέτο του γάλακτος, τα πρότυπα της ποιότητας, Παρακαλώ αγνοήστε τα, γιατί αυτά θα συζητηθούν ε, ξεχωριστά, βάσει ξεχωριστών προτάσεων που έχουν υποβληθεί. Τώρα, αν μπούμε και σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το πλαίσιο, τότε θα καθυστερήσουμε περαιτέρω την υιοθέτηση. Γι' αυτό προσπαθούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στο θέμα της ευθυγράμμισης. Σε αυτή τη βάση λοιπόν, Πρόεδρε, καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξάγει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον και τη Γενική Διευθύνση Γεωργίας για το έργο της. Μέσω του κυρίου Ογκάρτ ε, θέλουμε να στείλουμε και ένα ευχαριστώ στον Επίτροπο, γιατί όπως ακούσατε αυτή η εξισορρόπηση μεταξύ εκτελεστικών ε, πράξεων ε, και κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι μία οδός η οποία μας βρίσκει σύμφωνους αλλά και επιθυμούμε να ακολουθήσουμε και αυτή η αρχή της πρόληψης ε, στην οποία αναφερθήκατε Ελπίζω να μας οδηγήσει στο να δραματίσει το Κοινοβούλιο ένα ρόλο που ποτέ δεν θα το οδηγήσει στον παραγωνισμό. Έτσι λοιπόν εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να κινηθούμε όσο το δυνατόν συντομότερα και ελπίζουμε μέχρι τον Ιούνιο να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Οι ανησυχίες όμως που πρέπει να εκφράσουμε εδώ είναι ένα του Συμβουλίου. Φοβόμαστε ότι μπορεί να μην έχει βούληση να επιταχύνει στο χάκελο αυτό. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό, να επενδύσω συναδέλφους ε, ότι εδώ μιλάμε για τις εκτελεστικές πράξεις και για τις κατοξιδότητες πράξη. Κατοξιδότητες πράξη σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο συνεχίζει να δραματίσει ένα ρόλο και στην επακόλουθη συζήτηση ενώ στις εκτελεστικές πράξεις αποκλείεται το Κοινοβούλιο. Έτσι η επιλογή λοιπόν μεταξύ του ενός και του άλλου και αυτή, να υπάρχει αυτή η ισορροπία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και για μας σημαίνει ότι αν θα σεβαστούμε το πνεύμα της αγώνας ή αν δεν θα το σεβαστούμε. Έτσι λοιπόν εγώ είμαι πάρα πολύ μέσα από αυτή την παρουσίαση και μάλιστα και ο λόγος που οι συντονιστές αυτής της Επιτροπής διάλεξαν τις πρώτες εκτέσεις ε, ήταν και ο ίδιος που ασχοληθήκε για να δώσει μια κατευθυντηρία γραμμή που να μπορέσει να μας βοηθήσει για να κινηθούμε όσο δυνατόν συντομότερα έχοντας κατά νου ότι οι επόμενες μεταρρυθμίσεις θα έχουν αντίκτυπο και σε αυτή την επιλογή. Θέλω να υποστηρίξω τώρα ότι η βοήθεια που ζητάμε εμείς από την Κομισιόν έχει να κάνει με το να κινηθούμε ως το πιο γρήγορα γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να προκληθούν δυσκολίες από το Συμβούλιο που μάλλον θα είναι λιγότερο ενθουσιώδες για την ταχεία υιοθέτηση των πράξεων. Κλάς, έχετε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τονίσατε ότι συζητούμε αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρά θέματα. Σας ευχαριστώ για αυτό. Ευχαριστώ και τον κύριο Χόλκαρτ για την εισαγωγή που μας έκανε για το θέμα αυτό. Αλλά ε, μιλάμε για σοβαρά θέματα ε, αλλά έχω και κάποιες ανησυχίες. Φοβάμαι ότι δεν πρόκειται απλά για μια προσαρμογή στις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Φοβάμαι ότι ε, επιχειρούνται και πολύ περισσότερα πράγματα εδώ. Δεν πρόκειται απλώς για απλούστευση της ΚΑΠ και αυτό βεβαίως δεν θα έβρισκε αντίθετο κανένα ο κύριος Χόλκατ ε, είπε ότι βεβαίως το θέμα είναι τεράστιο ε, έχουν γίνει πολλές αλλαγές αναφέρθηκε στις αλλαγές που έγιναν για το κρασί και υπενθυμίζω ότι στην υπόθεση του εμπελονικού τομέα απλώς είχαν ζητηθεί κάποιες τελείως τεχνικές αναπροσαρμογές και όμως ε, και πιστεύω ότι ε, όπως και εκεί έγιναν παραπάνω από τις τεχνικές αναπροσαρμογές και εδώ επιχειρείται το ίδιο. Στην ημερήσια διάταξή μας, εκτός από το σημείο 3, έχουμε και το σημείο 4, που νομίζω είναι σχετικό. Και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α, ε, ξέρει, γνωρίζει τις α, ε, α, ε, καινούργιες προτάσεις για τις α, εκτελεστικές πράξεις, εφαρμοστικές πράξεις και τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και ακόμη και για τις κατα... και, για τις κατεξουσιοδότης πράξεις έχει το Κοινοβουλίο τη δυνατότητα να παρέμβει και βεβαίως έχει και την πολιτική ευθύνη να παρέμβει αν νομίζει ότι πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο και η Κομισιό μπορεί να θα μου πείτε ε, να έχει πολιτική ευθύνη αλλά εμείς σαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των λαών μας ε, πρέπει να ε, ε, πούμε ότι έχουμε την κύρια πολιτική ευθύνη εδώ και ε, Βεβαίω μα λέει ο κύριο Χόλκαρτ ότι έγιναν μελέτες, έγιναν πολλές σκέψεις, έγιναν πολλά πράγματα, προτείνονται πολλά πράγματα που είναι τελείως εξισορροπημένα. Ναι, αλλά αυτή την ισορροπία θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να την μελετήσουμε κι εμείς. Ε, αλλά τι να σας πω υπάρχουν θέματα παραδείγματο χάρη δημόσια αποθεματοποίηση ε, υπάρχουν θέματα στα οποία ενέχουν εμπλέκονται και χρηματοδότηση και ε, τα κράτη-μέλη βεβαίως ε, και ξέρω πολύ καλά ότι το Συμβούλιο ζητεί και αυτό να μπορεί να επέμβει και όχι μόνο εκ των υστέρων για να εκφράσει ενστάσεις αλλά ήδη από την αρχή για να μπορέσει να συνδιαμορφώσει ορισμένα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ και δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να πούμε ότι αφήνουμε να την Κομισιόν να κάνει τη δουλειά. Ε, εδώ πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχουν και κρεμούν ακόμη πολλά πράγματα. Ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας κύριε Κλάσπ αρχίζουμε τώρα να εξετάζουμε το κείμενο της Κομισιόν. Φυσικά θα προσπαθήσουμε και εμείς να πούμε την άποψή μας στη συζήτηση που θα έχουμε να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά εκθετική προσέγγιση της ε, της Γεωργίας και όσο μας είπε ο Ούκαρτ ε, και συγκεκριμένα για το άρθρο 43 παράγραφος 3. Φυσικά εκτιμήσαμε τόσα είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν θα ήταν καλύτερο να μην υπήρχε αυτό το άρθρο και αυτή η παράγραφος. Ε, δυστυχώς μας φέρνει αυτό σε δύσκολη θέση. Και καθώς το Συμβούλιο εδώ βάζει από το παράθυρο ότι έβγαλα την πόρτα. Αυτή η προσέγγιση θα παγιωθεί στο έργο που θα κάνουμε για την ενιακό. ΚΟΑ. Πάντως, ε, εκτιμήσαμε και στο ότι αυτή, σε αυτή την ε, ε έκθεση θα πρέπει ε, εδώ να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση να κάνουμε αλλαγές ε, ε, για νομοθεσία η οποία είναι υπό εκπόνηση. Θέλω να ζητήσω από τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν, να ρωτήσω τον εκπρόσωπο τη Κομισιόν αν θέλει να πάρει το λόγο να προσθέσει κάτι. Διαφορετικά, να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, απλά να δώσω ένα-δυο συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί όπως είπε και η κυρία Κλάς, ε, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα, μιλάμε για την αποθεματοποίηση, υπάρχουν πολλές πολιτικές προσεγγίσεις και τα λοιπά. Είναι δύσκολο και πρέπει να γίνεται κάποιος έλεγχος. Συμφωνώ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί αν θέλαμε να είμαστε τέλειοι θα έπρεπε κάθε μέρα να κουβεντιάζουμε τα θέματα αυτά. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό η αποστολή σας. Η αποστολή σας είναι να μπορείτε, αν υπάρχει κάποιο θέμα ευαίσθητο που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο, να μπορείτε να παρέμβετε, να παραμβαίνετε. Όταν μιλάμε λέει, για καταεξουσιοδότηση πράξης, ε, να μπορείτε να παρεμβαίνετε, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι η εξαίρεση. Εμείς σαν Κομισιόν ε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να είμαστε αρκετά ε, προσεκτικοί, να είμαστε αρκετά ε, για να, να κάνουμε τα πράγματα καλά αλλά εσείς θα πρέπει να επεμβαίνετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αλλά αυτό σε ε, σπάνιες περιπτώσεις και αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επικεντρώσετε την προσοχή σας στα ιδιαίτερα λεπτά και ευαίσθητα θέματα αλλά ο κανόνας πρέπει να είναι τα πράγματα συνεχίσουν να προχωρούν όπως μέχρι τώρα ε, μπορεί η Κανονιστική Επιτροπή, η τωρινή Ρυθμιστική Επιτροπή να αλλάξει. Δηλαδή δεν μιλάμε για επανάσταση, δεν μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν στο Κάιρο και την ε, ανατροπή του καθεστώτος. Μιλάμε για ε, πολύ πολύ πολύ μικρότερες αλλαγές. Λοιπόν, είπα θα σας δώσω παραδείγματα. Δείτε, πάρουμε την παρέμβαση, άρθρο 31. Στη σελίδα 56 της πρότασης, στο κείμενο 5084, όχι, λάθος, 2010 0385 της Κομισιόν. Λοιπόν, κοιτάζουμε τέλος πάντων το άρθρο 31. Ένα εδώ μιλάμε για κατεξουσιοδότηση πράξης και αναφέρονται οι όροι που πρέπει να πληρούνται από τα προϊόντα τα οποία μπαίνουν στην παρέμβαση. Στη δημόσια παρέμβαση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να ορίσουμε τις απαιτήσει ποιότητας για τα σιτηρά, ελάχιστο βάρος, τον αριθμό Χάγκμπεργκ, πτώσεις Χάγκμπεργκ κλπ. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές πολιτικές διαστάσεις εδώ γιατί άμα πούμε αλλά από εκεί και πέρα ε, τα θέματα είναι μάλλον τεχνικά. Αν πούμε ότι θέλουμε περιεκτικότητα πρωτεΐνης 14% τότε τα ε, στερά που θα βάλει στην παρέμβαση είναι ελάχιστα. Αυτό θα ήταν μια πολιτική διάσταση αν θέλετε. Αλλά δεν πρόκειται για τέτοιου είδους πράγματα. Πρόκειται για τεχνικές λεπτομέρειες τεχνικούς καθορισμούς. Και δεν μιλάμε τώρα για την εφαρμογή. Εναρμόνιση ουσιαστικά. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο, με όμορφο τρόπο ε, κάποιες διατάξεις, έτσι. Για την παρέμβαση να οριστούν ε, οι, τα τεστ και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το, να αποφασιστεί αν κάποιο προϊόν μπορεί να μπει στην παρέμβαση ή όχι. Δεν υπάρχει πολιτική διάσταση εδώ. Είναι πάρα πολύ μικρή η πολιτική διάσταση εδώ. Υπάρχουν και σημεία, στοιχεία εδώ με πολιτικές διαστάσεις, αλλά όχι τα περισσότερα. Εδώ κυρίως μιλούμε για εφαρμογή και δι ομοιόμορφη, θέλουμε να επιτευχθεί ομοιόμορφη εφαρμογή στην καθημερινότητα. Τώρα, το 43-3, τι να κάνουμε. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα ότι είναι κρίμα που μπήκε εδώ, αλλά βεβαίως θα είναι αντικείμενο ξεχωριστής πρότασης που θα έρθει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και τότε θα, όταν θα υποβληθεί αυτή η ξεχωριστή πρόταση θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια ξεχωριστή συζήτηση βεβαίως και ελπίζουμε να συμφωνήσετε αλλά γι' αυτό το θέμα η συζήτηση δεν είναι κατά κύριο λόγο με την Κομισιόν κατά κύριο λόγο με το Συμβούλιο ναι, συμφωνούμε μαζί σας. Σας αναφέρω εδώ ένα κοινότυπο παράδειγμα, αλλά μπορούμε όλοι να εκτιμήσουμε εμείς την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε την πρόταση του Συμβουλίου για την παρέμβαση για την κρίση των χείρων. Είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο θέμα και θέλουμε στο μέλλον να έχουμε μια πράξη μέσα της οποίας θα μπορέσει να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο. Όμως ε, για, φυσικά για τα θέματα της πρακτικής εφαρμογής δεν θέλει το Κοινοβούλιο ε, να ε, καθυστερήσει τη διαδικασία της εκτέλεσης των πράξεων. Έτσι λοιπόν, ε, ξεκινάμε μια καλή βάση, θέλουμε να προχωρήσουμε το δυνατόν συντομότερο και ζητάμε τη βοήθεια της Κομισιόν για να, προωθεί, για να οθήσει το Συμβούλιο να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, σας περάσουμε και στο σημείο 4 που είναι παρόμοιο. Θέλω να χαιρετήσω το διευθυντή που είναι εδώ μαζί μα. Θα μιλήσουμε για την τροπήση του κανονισμου 1992. 1092-2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση τη κοινή γεωργική πολιτική και την κατάργηση των κανονισμών 165-94 και 78-2008 του Συμβουλίου. Αυτή είναι μια έκθεση την οποία έχει αναλάβει η ομάδα του ΕΛΚ, ακόμη δεν έχει όμως διοριστεί ο συγητής. Γι' αυτό θα δώσω απευθείας το λόγο στον Διευθυντή Λόγκο. Θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε, γιατί ο κύριος Σούγκαρτ ε, παρουσίασε με πολύ λιρότητα το ζήτημα, έτσι λοιπόν θα ήταν δύσκολο να προσθέσω κάτι άλλο, πέρα από το να πω κάτι ουσιαστικό που είναι το εξής, ε, ότι οι γραμμές καθορισμού που εμείς ε, χρησιμοποιήσαμε για τη διαφοροποίηση των δύο πράξεων, εκτελεστικών πράξεων και κατεξοδότηση πράξεων, εμπνέονται από τις ίδιες αρχές που ενέπνευσαν και την προηγούμενη πρόταση. Λεχθέντος αυτό μου φαίνεται ότι είναι δύσκολο. Να επανελθώ τουλάχιστον όχι με την ίδια επιτυχία που ε, παρουσίασε ο κ. Σούγκαρτ ε, την ε, προηγούμενη μεθοδολογία. Θα ήθελα λοιπόν απλώς να περιοριστώ στο να επισημάνω ένα στοιχείο που αναφέρατε κι εσείς δηλαδή την ε, ευκαιρία της ευθυγράμμισης, την οποία την αδράτουμε εμείς, και για να επιδιορθώσουμε κάποια γλωσσικά προβλήματα που υπήρχαν ε, σε αυτόν τον κανονισμό. Δηλαδή να βάλουμε μια τάξη, χωρίς να αλλάζουμε ουσιαστικά στοιχεία. Έχουμε τον ε, κανονισμό 78 του 2008 και τον 165 του 1994 ε, εντάσσουμε τα άρθρα 1 και 2 στη δική μας πρόταση κανονισμού. Λεφθαντός αυτό λοιπόν, πιστεύω ότι θα γλιτώσουμε χρόνο, Πρόεδρε, αν εγώ περιοριστώ. Εδώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Διευθύντα. Τζοβάνι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βλέπουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η Κομισιόν ξεκινά μια διαδικασία πλούστευσης των ευθυγραμμίσεων και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ότι στη διαδικασία της ευθυγράμμισης ε, επιζητούμε να μειώσουμε την πολυπλοκότητα της κοινωτικής νομοθεσίας. Ε, αυτό είναι σίγουρα κάτι θετικό. Και πιστεύω ότι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσει. Σε σχέση τώρα με το περιεχόμενο της ευθυγράμμισης, πιστεύω ότι η συζήτηση που έγινε προηγουμένω θα μπορούσε σε ένα μεγάλο βαθμό να αναπαραχθεί πιστά. Και σε αυτή την περίπτωση, για να μην μακρηγορούμε και χάνουμε χρόνο, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πράξουμε. Απλώς ε, θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Πιστεύω ότι η διαδρομή της ευθυγράμμισης θα πρέπει να καταστήσει πιο ταχύα τη διαδικασία της διαδικασίες μάλλον χωρίς ε, να υπάρχει γραφειοκρατία αφήνοντας ταυτόχρονα και στο Κοινοβούλιο την αυτονομία να διαδραματίσει ρόλο και υποβολής προτάσεων αλλά και ελέγχου και εγώ νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν κάποια βήματα ακόμη. Πιστεύω ότι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο γενικά θα, μάλλον και η Επιτροπή θα είναι σε θέση και θα είναι διαθέσιμε να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για αυτή την πρόταση ευθυγράμμισης. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλα. Κοιτάξτε, ε, θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία παραδείγματα εδώ. Στο άρθρο 35α λέγεται για να διορθωθούν ε, τα νούμερα των... για να διορθωθούν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει τα, ε, στοιχεία που έχουν δώσει τα κράτη-μέλη η Κομισιόν βάσει του 42α ε, θέτει ή επιβάλλει μάλλον τους κανόνες συμψηφισμού. Αυτά τα κάνει η Κομισιόν μόνη της στο 37α για να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή μπορεί η Κομισιόν σε μια κατεξουσιοδότηση πράξη να ορίσει διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις συνεργασίας των κρατών μελών και μόνη της Κομισιόν τα κάνει αυτά και στο άρθρο 40 3 λέγεται ότι η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει διατάξει για την περικοπή των πληρωμών στα κράτη-μέλη. Να, τρία παραδείγματα που κατά την άποψή μας ε, έχουν σοβαρές πολιτικές διατάξεις, Και παρακάτω στο άρθρο 42 της, ε, ε, του κειμένου λέγεται για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ότι οι πράξεις αυτές μπορούν να δημοσιευθούν στην ε, στην ε, επίσημη εφημερίδα πριν να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Γιατί όμως δεν αναφέρεται πουθενά ότι θα πρέπει εκ να γνωστοποιηθούν αυτές οι πράξεις για να ενημερωθεί ο κόσμος, να ενημερωθούμε εμείς, να ενημερωθούν τα κράτη-μέλη τις που έρχονται. Ωραία, αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Λόγκο. Αλλά ήθελα και εγώ να σας ε, καθησυχάσω. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε και ε, φυσικά να δεκτούμε αυτές τις αλλαγές. Ε, ξέρετε ότι θα έρθει και θα αντιταχθεί η Κομισιόν. Κύριος Λόγκο, θέλω να πω, Πρόεδρε, ότι πολλοί από αυτού του κανόνε, στους οποίους αναφερθήκατε είναι οι φυστάμενοι κανόνες. Υπάρχουν στη σημερινή νομοθεσία. Εμείς απλώς κάναμε μία μεταφορά, αλλά λειτουργώντας με τον ίδιο τρόπο όπως έχουμε λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Εδώ λαμβάνω υπόψη την πρόταση να εξετάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή ορισμένα σημεία ανησυχία στους αξιότιμους και τους βουλευτές. Και φυσικά είμαι διαθετημένος να συνεργαστούμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες ε, και απόψεις για τα θέματα αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν, κύριοι βουλευτές, ε, αν θέλετε να παρέμβετε σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και την Κομισιόν, ευχαριστώ τον Κρατ και τον Λόγκο. Και ας περάσουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, πολύ σημαντικό σημείο. Προσοχή λοιπόν. Τροποποίηση τη οδηγια 2018 σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροπομένων οργανισμών στην επικρατειά του. Ε, η συγητή είναι ο κ. Λάιον. Όπως όλοι γνωρίζουμε, πρόκειται για ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Πάντα προκαλεί ιδεολογικές συζητήσει και είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε την πρόταση της Επιτροπής με ρεαλιστικό τρόπο, έχοντα κατά νου ότι το Συμβούλιο ήδη έχει εκφράσει προβληματισμό επί της πρότασης αυτής. Πριν να δώσω το λόγο στον Τζόρτς, να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών έχει λάβει παράταση μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου. Έχουμε λοιπόν κάποιες μέρες ακόμη στη διάθεσή μας. Προθεσμία λοιπόν κατάθεση τροπολογίων 9 Φεβρουαρίου. George, έχεις το λόγο. Uh, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως πολύ σωστά είπατε, το ζήτημα αυτό δεν θα οδηγήσει εύκολα σε συνένεση ούτε σε κατάσταση αρμονίας. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το συζητήσουμε και θα πρέπει να το δούμε στα σωστά πλαίσια του. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για ανθρώπους που είναι υπέρ ή κατά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Γίνεται απλώς μια συγκεκριμένη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέψει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφος τους αν θα πρέπει να τροποποιηθεί, να ενδυναμωθεί η πρόταση αυτή. Είχαμε γνωμοδοτήσει από το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν τελικά υπάρχει μια νομική βάση για κάτι τέτοιο, για μια τέτοια πρόταση. Η νομική άποψη του Συμβουλίου είναι αρνητική, το Κοινοβούλιο στην νομική του γνωμοδότηση είπε ναι, αλλά κατά τρόπο ιδιαίτερα περιορισμένο και ανάλογη φαίνεται να είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίθεται ένα πολιτικό ζήτημα για την Επιτροπή μας. Είχα και συζητήσεις με τους σκιώδεις, τους έθεσα κάποιες ερωτήσεις. Ήθελα να δω αν θέλουν να απορρίψουμε την πρόταση αυτή. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε καθόλου, γιατί από ό,τι φαίνεται η Επιτροπή περιβάλλοντος δεν θα μας ακολουθήσει ή θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εδώ πέρα στη συζήτηση και την ε, οπτική γωνία των γεωργών των ε, καλλιεργητών. Και οι περισσότεροι με μία ουσιαστικά εξαίρεση είπαν ότι θα πρέπει να εμπλακούμε και εμείς στη συζήτηση και να προχωρήσουμε με αυτή την πρόταση. Αυτό προσπάθησα λοιπόν να κάνω είναι κοιτάζοντας όλες τις εναλλακτικές λύσεις και προσπαθώντας να δυναμώσω τελικά την πρότασή μας αυτή, λέμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν ληφθούν όμως υπόψη πρώτε τροπολογίες και αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Δεχόμαστε την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πρόταση αυτή ενδεχομένως να πετύχει τους στόχους της, δηλαδή να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία και να βρωθεί μια λύση στο υφιστάμενο αδιέξτο που υπάρχει με την αδειοδότηση για την καλλιέργεια αυτών των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Προσπάθησα επίσης να δω πώς θα μπορούμε να προστατεύσουμε οικονομικά τους καλλιεργητές μη γενετικά τροπημένων ε, φυτών, οργανισμών και πώς ε, μπορούμε να διευθετήσουμε και τις επιθυμίες κάποιων κρατών ή περιφερειών που σε τοπικό επίπεδο θέλουν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια αυτών των ε, οργανισμών, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Το σημείο κίνησης ήταν μάλλον μια βασική αλλαγή που έχει γίνει είναι ότι έχουμε την αρχή της αναλογικότητας, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλέον τα κράτη-μέλη. Επίσης, λέγεται επίσης ότι θα μπορούσε να γίνει μια διαδότηση βάσει συγκεκριμένων φυτών, συγκεκριμένων καλλιεργειών, γιατί από τη μία καλλιέργεια στην άλλη επίδραση στο περιβάλλον περιβάλλον μπορεί να είναι εντελώ διαφορετική. Θέλουμε επίσης να δούμε αν τίθεται κίνδυνος από κάποιες συγκεκριμένε καλλιέργειες, πώς μέσω της γύρης θα μπορούσαν ενδεχομένως οι γενικά τροποποιημένοι οργανισμοί να μεταφερθούν και σε άλλες καλλιέργειες και πώς μπορεί να αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει ένα ευέλικτο σύστημα ελεύθερης επιλογής, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση με βάση την καλλιέργεια, κατά περίπτωση καλλιέργεια δηλαδή. Επίσης έχουμε και το άρθρο 26 και την ε, δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ακόμα και η απαγόρευση ως ε, έσχατη λύση. Και επίσης προβλέπονται και κάποια μέτρα συνύπαρξης στο άρθρο 26α αντί να λέμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θετήσουν μέτρα συνύπαρξης, λέμε ότι θα υιοθετήσουν μέτρα συνύπαρξης. Χρησιμοποιείται η λέξη shall στα αγγλικά, στο αγγλικό κείμενο. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται και η ενδεχομένως ανάμιξη, η ανάμιξη που θα μπορούσε να προκύψει στους σπόρους και η οποία θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις. Υπάρχει βέβαια και αρχή αναλογικότητας, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, αναφερόμαστε και σε μια άλλη αρχή, ελεύθερη επιλογή τόσο των γεωργών όσο όμως και των καταναλωτών. Οι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την επιλογή, το ίδιο όμως θα πρέπει να μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι οι καταναλωτές. Και περνάμε στο πέμπτο σημείο, όπου ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε ένα κατώτατο όριο τεχνικό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει προκειμένου να προστατευθούν οι γεωργοί αυτοί οι οποίοι δεν καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ορισμένοι λένε ότι το όριο αυτό θα πρέπει να είναι μηδενικό, να μην υπάρχει δηλαδή καμία δυνατότητα μόλυνσης. Αν όμως δούμε οποιασδήποτε άλλες πολιτικές κατά της μόλυνσης, είτε πρόκειται για το νερό, είτε πρόκειται για τη διοξίνη, έχουν τεθεί από, τις, από τους αρμόδιους φορείς τέτοιες, ε, τέτοια κατώτατα όρια. Πολλές φορές δεν μπορούμε να έχουμε την αυτή, ε, το μηδεμινό αυτό περιθώριο. Επομένω, θα πρέπει μια ανάλογη αρχή να ακολουθηθεί και εδώ προκειμένου να μπορεί να ισχύει η ελεύθερη επιλογή και για τους καλλιεργητές από τροποποιημένων οργανισμών και για αυτούς που δεν δέχονται να καλλιεργήσουν τέτοια φυτά και για τους καταναλωτές. Επίσης, ε, ζήτησε και μια γνωμοδότηση για την ε, νομική ασφάλεια για τους ε, γεωργούς εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να καλλιεργήσουν γενικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να ενημερώνονται οι γεωργοί αυτοί τρεις μήνες πριν ξεκινήσει η καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών από άλλους γεωργούς, προκειμένου να δίνεται και δυνατότητα σε κυβερνήσεις ή τοπικές κυβερνήσεις να, λαμβάνουν μέτρα απαγόρευσης. Ορισμένοι πρότειναν να έχουμε έναν κατάλογο με συγκεκριμένα εδάφιο που θα μάλλον τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, οι διατάξεις αυτές. Εγώ είπα ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κατέληγε σε έναν μη εξαντλητικό κατάλογο τους ή άλλως. Επίσης, ε, εναπόκειται πολλές φορές στα αρμόδια δικαστήρια να αποφασίσουν αν οι λόγοι αυτή αδειοδότηση είναι έγκυροι ή όχι. Επομένω, δεν υπήρχε λόγος να καταρτιστεί από την Επιτροπή Κατάλογος, ο οποίος δεν θα ήταν διεξοδικός. Πιστεύω επίσης ότι το ζήτημα το περιβαλλοντικό και της προστασία προστασίας της υγείας δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτή τη στιγμή στη διαδικασία που εμεί ακολουθούμε, γιατί διαφορετικά θα καταλήξουμε σε 27 διαφορετικέ ερμηνείε ή σε εκατοντάδε διαφορετικέ ερμηνείε, αν συμπεριλάβουμε και τι τοπικέ κυβερνήσει. Στο να πούνε δηλαδή και αυτέ τι είναι ασφαλέ και τι δεν είναι, ή τι είναι φιλοπεριβαλλοντικό, τι δεν είναι. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο και δεν θα καταφέρναμε τελικά να επιτελέσουμε σωστά το στόχο μας εδώ πέρα, που είναι η προστασία τόσο των γεωργών όσο και των καταναλωτών όσον αφορά τα προϊόντα. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν, να ενδυναμωθούν λίγο περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό πάντως το σύστημα αδειοδότησης και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την ασφάλεια του περιβάλλοντος ή για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας να είναι κοινέ, να βρίσκονται δηλαδή να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν θα πρέπει οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία να βάλλονται από διαφορετικές ερμηνείες που μπορεί να υπάρχουν από τη μία χώρα στην άλλη. Έκανα λοιπόν κάποιες σχετικές τροπολογίες η Επιτροπή περιβάλλοντο είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή σαφώ. Αυτοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ σημαντικό όμω και εμεί να καταφέρουμε να υποβάλουμε τις δικές μας προτάσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και θα μας δοθεί και η δυνατότητα να υποβάλουμε και νέες τροπολογίες στην Ολομέλεια, να αυτό κρυθεί αναγκαίο. Είπατε κύριε Πρόεδρε ότι θα έχουμε ε, προθεσμία μέχρι την 9η Φεβρουαρίου για να υποβληθούν τροπολογίε. Η τελική ψηφοφορία επίσης θα θέλαμε να μην γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, είναι μια Δευτέρα μετά από μια πράσινη εβδομάδα και νομίζω ότι είναι δύσκολη η ημερομηνία αυτή, ιδίω αν λάβουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Θα είναι δύσκολο να τις συντάξουμε ουσιαστικά, να καταλήξουμε στις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Και εγώ και οι σκιώδες λοιπόν οι εισηγητέ θα θέλαμε να πάμε μια εβδομάδα μετά. Υπάρχει ε, ένα περιθώριο τριών εβδομάδων στη συνέχεια για την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να υποβάλουν τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να δοθεί και σε εμά μία επιπλέον εβδομάδα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρω να ακούσουν και τη δική μας την άποψη, προτού προχωρήσουν και αυτοί, οι συνάδελφοι δηλαδή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην δική τους τελική ψηφοφορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και συγητές για την καλή συνεργασία που είχα μαζί τους μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ, Τζόρτζ. Βεβαίω θα αναβάλουμε την ψηφορία για 15 Μαρτίου. 15 Μαρτίου, λοιπόν. Δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να πάρουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε. Αν λάβουμε υπόψη και τις ε, δύσκολες σχέσεις που έχουμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή Περιβάλλοντος επέμεινε στη συνεδρίαση των συντονιστών να ζητήσει την εφαρμογή του άρθρου 50 για την ΚΑΠ. Έτσι λοιπόν δεν θέλει να εκφράσει η γνωμοδότηση, αλλά θέλει να συναποφασίσει μαζί μα ε, για την κοινή αγροτική πολιτική. Εμεί είμαστε αντίθετοι, προετοιμάζουμε ένα σημείο για όλου του ηγητέ και έδρα την ευκαιρία να το ξαναπώ και εδώ. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη δική μα επιτροπή. Έτσι λοιπόν θα ψηφίσουμε στις 15 Μαρτίου για του γάμματα αφόμικρων. Λοιπόν, να δώσω τον λόγο στον Αντιπρόεδρο Νικολάσικο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάιον για το σχέδιο γνωμοδότηση που μας παρουσίασε. Είμαι πεπισμένος ότι ε, δεν ήταν εύκολο. Επρόκειτο για ένα λεπτό ζήτημα. Θα ήθελα επίση ε, να τονίσω το ρεαλισμό της ε, γνωμοδότησης. Ε, πιστεύω ότι εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική που να ευνοεί τους καταναλωτές και τους γεωργούς. Και αυτό μας ε, προτείνει η γνωμοδότηση, αλλά και οι τροπολογίες του Τζόρτς. Και, όπως είπε και ο συντάκ, της γνωμοδότησης περιλαμβάνονται εδώ και τα θέματα της επικουρικότητας. Μία από τις τροπολογίες που διάβασα με οδηγεί στο να σκεφτώ ότι δεν ξέρω ποια είναι η διαφοροποίηση μεταξύ της τροποποίησης που προτείνει ο εισηγητής ό,τι αφορά τα μέτρα απαγόρευσης γενετικά τροπημένων οργανισμών ανά περίπτωση ποια είναι η διαφορά της δική τους πρότασης σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Πάντως όπως και να έχει είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αυτή η πρωτοβουλία αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε και εμείς εδώ παραδείγματο χάρη τη λύση που θα δοθεί για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών καθώς ε, πολλές φορές ε, είναι ένα θέμα που είναι δύσκολο να, το εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας. Ο κύριος Μπουβέ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάιον. Άκουσα αυτόν τον απολογισμό που κάνατε, την εργασία την οποία επιτελέσατε με τους κοιόδης εισηγητές και βλέπουμε και ποιο είναι και το σχέδιο το οποίο προτείνεται μετά το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε από την αρχή την όλη συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Ας είμαστε όμως συγκεκριμένοι. Θα κάνω ένα πρώτο σχόλιο. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι έχουμε μια πλειονότητα, μια πλειοψηφία κρατών μελών που δεν θέλει την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν προσθέσουμε και τα κράτη-μέλη που απέχουν, έχουμε ένα τρίτο περίπου των κρατών μελών. Επίσης, Έχουμε και μια ολόκληρη συζήτηση για τα οικονομικά πρότυπα, τα οποία επιβάλλονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τα όσα ισχύουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί πρόβλημα. Τρίτον τώρα. Όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσέχει και την κοινή γνώμη. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη σήμερα. Και μάλιστα έχουμε 1.500.000 άτομα που υπέγραψαν μία αίτηση και την οποία υπέβαλαν μάλιστα στον Επίτροπο Ντάλι προκειμένου να σταματήσει η καλλιέργεια γενετικά τροπημένων οργανισμών. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η πραγματικότητα σε πάρα πολλές περιφέρειες της Ευρώπης και έχουμε και πολλούς ευρωβουλευτές εδώ που προέρχονται από περιφέρειες που υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των πολιτών. Ας προσέξουμε λοιπόν να μην βρισκόμαστε εμείς σε εντελώς διαφορετική φάση και τόνο από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πράξη, από αυτά τα οποία ζητούν οι πολίτες. Θα ήθελα συγκεκριμένα να αφαιρθώ τώρα στις προτάσεις σας και θα ήθελα να σας δείξω ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με τους σπόρους. Στην τροπολογία σας 4 στο εκτιμώντας 8 λέτε ότι θα πρέπει σε σχέση με τους σπόρους να αναφερθούμε σε ένα κάποιο κατόφλι, ότι μπορεί να υπάρχει ένα κάποιο ανεκτό όριο για γεννητικά τροπημένους οργανισμούς. Αυτό το κατόφλι σήμερα είναι μηδενικό. Είπατε βέβαια εσείς ότι υπάρχουν άλλα κατόφλια τα οποία δεν είναι μηδενικά για τα ζενεοκτώνα κτλ. Ουσιαστικά όμω δεν συνειδητοποιείται το πέρα τη κατάσταση, γιατί αν για ένα χρόνο δεχτούμε 0,3%, τον επόμενο χρόνο θα έχουμε αναγκαστικά μία αύξηση και θα πάμε στο 0,8 ή στο 1% και μετά θα πάμε στο 3 ή στο 4% και θα φτάσει η στιγμή εκείνη που θα είναι αδύνατο να έχουμε πλέον σπόρους οι οποίοι θα είναι καθαροί 100% χωρί γενετικά τροπημένου οργανισμού. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί λοιπόν ω προς τους σπόρους. Είτε θα έχουν γενετικά τροπημένου οργανισμού, είτε δεν θα έχουν. Δεν μπορούμε εδώ πέρα να επιτρέψουμε την βαθμία αυτή μόλυνση των σπόρων από του γεωργού αυτού οι οποίοι δεν θα σέβονται τις ε, ζώνες εκείνες ε, σποράς καταλαβαίνετε ότι αν ξεκινήσει μία μόλυνση στους σπόρους, σιγά σιγά αυτή θα αυξηθεί, αναγκαστικά, εκ των πραγμάτων. Δεύτερον τώρα σημείο στο κείμενό σας με το οποίο έχω πρόβλημα, Νομίζω ότι δεν είναι ρεαλιστική αυτή η χρονική περίοδος των τριών μηνών για να εφαρμοστεί μια πολιτική. Γιατί όταν μπούμε στη διαδικασία αυτή βλέπουμε ότι ε, τους σπόρους αυτούς τουλάχιστον έξι μήνες εκ των προτέρων αρχίζουν και τους διαχειρίζονται οι μεγάλες αυτές εταιρείες και ξέρουμε ότι ε, για τον Αραβόσιτο για παράδειγμα οι αγορές που γίνονται από τους γεωργούς, οι παραγγελίες γίνονται τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο προκειμένου τέλη Απριλίου ή Μάιο να, γίνει, να φυτευτούν οι σπόροι αυτοί. Αν λοιπόν πάρουμε μόνο τη φάση αυτή που επιλέγει ο Γεωργός, τότε θα πρέπει να προβλέψουμε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Διαφορετικά η προσέγγιση μας δεν είναι ρεαλιστική. Τρίτον, το είπατε κι εσείς, όλο αυτό το ζήτημα των μέτρων συνύπαρξης. Πώς μπορούμε να οργανώσουμε αυτή την συνύπαρξη. Λέτε ότι θα πρέπει να ενδυναμωθούν τα μέτρα συνύπαρξης. Αν δείτε όμως τον αριθμό των κρατών που σήμερα έχουν εγκρίνει μια κάποια νομοθεσία συνύπαρξης, αν δεν κάνω λάθος είναι ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε το πολύ χώρες. Γιατί στην πράξη τίποτα δεν έχει γίνει. Στη Γαλλία για παράδειγμα, στη δικιά μου τη χώρα, έγινε μια τεράστια συζήτηση. Ψηφίσαμε νόμους, αλλά οι νόμοι αυτοί δεν έχουν εφαρμοστεί γιατί δεν έχουν εγκριθεί συγκεκριμένοι κανόνες. Το να βασιστείτε λοιπόν σε αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Την ημέρα που θα έχουμε όλα τα κράτη-μέλη που θα έχουν εγκρίνει τέτοιου συγκεκριμένου κανόνε, τότε ναι, α κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγο. Και τελευταία παρατήρηση. Θα ήθελα να αφαιρθώ στον κατάλογο εκείνων των λόγων άρνησης της καλλιέργειας. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε κάποια επιστημονικά δεδομένα, πραγματικά επιστημονικά δεδομένα, αναλυφθούν υπόψη και κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί, οικονομικοί παράγοντες, γιατί οι επιπτώσεις είναι πάντα σφαιρικές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να, να αναφερθούμε στο σύνολο των ζητημάτων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay, no. Ωραία. Ο κύριος Σενιού και κατόπιν Λόσοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε το πώς, πότε και πώς μπορούν να καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο θέμα που συζητιέται επί χρόνια, τίποτα δεν έχει συμβεί, πλήρης παράλυσης, υπάρχουν βεβαίως επιστημονικά δεδομένα. Στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο η υπάρχουν διστάμενες απόψεις ε, κάποιοι είναι καλλιεργούμε βέβαια κάποιοι γενετικούς ε, τροποποιημένους οργανισμούς αλλά υπάρχουν μερικοί που είναι υπέρ μερικοί που είναι κατά εγώ νομίζω ότι η απόφαση θα πρέπει να περθεί από τους πολίτες της χώρας μας και όχι από την Επιτροπή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε λέει ο κύριος Βλόσοβιτς Κυρίες και κύριοι, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, το θέμα είναι δύσκολο. Το οποίο συζητιέται βέβαια πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να παρθούν κάποιες σαφείς αποφάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τα κράτη-μέλη Βεβαίως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουν αρκετό περιθώριο για να αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να καλλιεργήσουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αλλά υπάρχουν πολλές διστάμενες απόψεις και αμφιβολίες ακόμη και από την νομική υπηρεσία του, του Κοινοβουλίου. Το... Εγώ νομίζω ότι ένας γενικός στόχος για τη δημιουργία νέων ευκαιριών για ορισμένους ή για ορισμένες ε, χώρες δεν είναι ένας στόχος το, με τον οποίο είναι τόσο φλού στόχος δεν αξίζει να ασχοληθούμε. Θα πρέπει να μπορούν τα διάφορα κράτη-μέλη να αποφασίζουν εάν θέλουν να καλλιεργούν τέτοιους οργανισμούς ή όχι και ο κανονισμός αυτός ακόμη και αν ο τίτλος του είναι σαφής ε, τελικά θα παραμείνει νεκρό γράμμα γιατί διότι φοβάμαι ότι δεν θα έχουν τα απαραίτητα εργαλεία τα κράτη-μέλη για να εφαρμόσουν τον κανονισμό αυτό ο κύριος Κόστιντζερ κυρία Κόστιντζερ ευχαριστώ πρόεδρε Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε και πραγματικά χαιρετίζω το γεγονός ότι καταρχήν ο εισηγητής δέχεται την πρόταση της Κομισιόν και λέει και αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ο δικαίωμα επιλογής το από πλευράς διαφόρων κρατών μελών. Ε, ετέθη ήδη το θέμα των σπόρων ε, η εισαγωγή όχι σπόρων από τρίτες χώρες και ποιών σπόρων Βεβαίω θα πρέπει να αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από εκεί και πέρα στα διάφορα κράτη-μέλη η έγκριση όχι. Θα πρέπει να δίνεται με μια διαδικασία πιο διαφανή από ό,τι αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν, έχουν τα τεθεί η τροπολογίες που έχουν σαν στόχο τη διευκρίνηση της πρότασης της Κομισιόν ε, φοβούμε ότι θα υπάρχουν και άλλες τροπολογίες δεν μπορώ ο τέλος να συμφωνήσω με τον εισηγητή που λέει ότι ε, θέματα που άπτονται της δημόσιες υγείας και υγειονομικών ε, θεμάτων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για, την, για το θέμα που συζητούμε. Λάθος. Ε, ίσα ίσα εγώ νομίζω ότι πολύ σημαντικό επιχειρήματα για να πάρθει η τελική απόφαση υπέρ κατά κάποιου γενετικά τροποποιημένου οργανισμού είναι το θέμα της δημόσιας υγείας. Επίσης, τα, αυτό που λέγεται εδώ ότι τα κράτη-μέλη θα τα κράτη-μέλη μπορούν κατά περίπτωση να αποφασίζουν έτσι όπως αναφέρεται αυτό εδώ δεν με βρίσκει σύμφωνη διότι αυτό περιορίζει την ελευθερία επιλογής των κρατών μελών νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να είναι απολύτως ελεύθερα ε, να διαλέξουν και τη μέθοδο με την οποία προχωρούν στην απαγόρευση όχι της καλλιεργίας κάποιων οργανισμών. Ο εισηγητής είπε ότι ε, ορισμένες τροπολογίες ε, θα έκαναν πολύ πιο αυστηρό αν θέλετε το κείμενο ε, ιδιαίτερα σε σχέση με τους ε, σπόρους υπάρχουν και κάποιες νομικές πτυχές εδώ που ε, δεν θα πρέπει να αγνοηθούν όπως παραδείγματος χάνει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για κάποιους σπόρους αυτά είναι πράγματι σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει ακόμη να δούμε και είμαι πεπισμένη ότι θα γίνουν ακόμη πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό η για τη συνύπαρξη τώρα ε, η, δεν αμφισβητώ ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να καλέσουμε την Κομισιόν να κάνει ε, να, να ετοιμάσει μία τεχνική ακόμη πιο λεπτομερή πρόταση για το θέμα αυτό ξεχωριστή αγαπητοί συνάδελφοι ε, ξέρουμε ότι στο Συμβούλιο ε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και θα συνεχίσουν να γίνονται συζητήσεις. Όμως στο Συμβούλιο υπάρχει ο φόβος της ανάληψης πολιτικής ευθύνης. Εμείς δεν έχουμε το φόβο αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε την απόψή μας. Ο κύριος ε, Μάρτιν Πρόεδρε, μετά από αυτά που είπαν οι προηγούμενοι δεν έχω πολλά πράγματα να πω ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση του Μποβέ τι να πω σίγουρα ε, ε αυτές είναι πολύ σημαντικές αποφάσεις οι διάφορες πολιτικές ομάδες ε, πρέπει να πάρουν θέση ένα όμως ένα είναι θέμα θα θέλω να αναφέρω γιατί δου, εμείς που είμαστε κατά των α, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ε, επικρινόμαστε πολύ συχνά ότι είμαστε μόνο συναισθηματικοί στις προσεγγίσεις μας και ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία τα οποία δεν ε, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ε, αυτό που υποστηρίζουμε και εμείς και είμαστε κατά αυτών των οργανισμών. Λάθος, διότι το ένα εκατομμύριο υπογραφές που συνελέγησαν νομίζω δείχνει ότι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και κύριε George Lyon, ε, έχω την εντύπωση ότι κάπου ε, κάποιοι προσπαθούν ή οι φιλελεύθεροι μάλλον προσπαθούν να βρουν ενδιάμεσες λύσεις ώστε να ε, καταργηθεί αν θέλετε το δόγμα της μηδενικής ανοχής που υποστηρίζουν ορισμένοι και, και εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό πράγματι δεν έχουν νόημα τα κατόφλια αυτά το 01, 03 και δεν ξέρω τι άλλο επιμόλυνση ουσιαστικά των σπόρων δεν εμείς είμαστε υποστηρίζουμε την αρχή της μηδενικής ανοχής και αυτό πραγματικά πρέπει να το τονίσουμε. Επίσης κάτι άλλο μου δημιουργεί αμφιβολίες, αν όχι υποψίες. Η τροπολογία περιθμών 5 για τη συνύπαρξη που λέει ότι ουσιαστικά για να ε, α, διευκολυνθούν ορισμένα πράγματα και αναφέρεται και η επαναθηνικοποίηση εδώ. Τι είναι δηλαδή αυτό. Συγγνώμη είναι άλλος φόβος αυτός που μας διακατέχει και περιγράφεται εδώ. Τα κράτη-μέλη παίρνουν κάποιες αποφάσεις αλλά μετά θα μπορούσαν για κάποιους λόγους να επαναχωρήσουν σε σχέση με τις αποφάσεις αυτές. Δεν μπορώ να καταλάβω περί τίνος πρόκειται εδώ. Και σε τελευταία ανάλυση, σε τελευταία ανάλυση εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους οργανισμούς αυτούς τι θα κάνουν θα τους επιβαρύνουμε με επιπλέον κόστη από εδώ και από εκεί έχουμε μια κοινή αγορά ή όχι διότι κάτι τέτοιο νομίζω ότι ε, υπονοείται εδώ τα κόντι δαπάνε των ελέγχων, πώς μοιράζονται κτλ. Όχι. Ε, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Βεβαίως θα υπάρχουν νομικά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν αλλά αυτές τις ακραίες θέσεις της αν θέλετε κατά αυτόν που είναι ενάντια στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν μπορούμε να το δεχθούμε και αυτά επιχειρήματα για τον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό του ε, Εμπορίου και τα λοιπά επίσης δεν μπορώ να τα δεχτώ Ρούμπιξ και μετά ο κύριος Σμιτ Ευχαριστώ πρόεδρε Άκουσα πολύ προσεκτικά τον εισηγητή και μπορώ να συμφωνήσω μαζί του. Λαμβάνοντα υπόψη τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε συνήθω όλα αυτά τα στοιχεία και διεξάγουμε τι συζητήσει. Και λαμβάνοντα υπόψη τα όσα λένε οι παραγωγοί. Η περισσότερη παραγωγή είναι υπέρ της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη χώρα μου δηλαδή. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι δημοκρατική εφόσον δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποιες ε, συστάσεις και αναφέρεται σε ένα 3% των τοπικών, ε, της ατοπικής αυτοδιοίκησης που ρυθμίζουν την ε, παραγωγή καλλιέργεια γενικά τροπημένων οργανισμών. Δεν έχουμε δει λοιπόν συγκεκριμένα προβλήματα με την εφαρμογή του συστήματο αυτού. Άκουσα και του συναδέλφου αυτού, οι οποίοι θέλουν να, έχουν πιο αυστηρού κανόνε και περισσότερου περιορισμού. Ω προ αυτό πιστεύω ότι μέχρι να καταλήξουμε στελικά αποτελέσματα θα έχουμε και τη δυνατότητα να εξετάσουμε την κατάσταση καλύτερα, να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό. Συμφωνώ πάντως. Ευχαριστώ. Smith. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι... Συγγνώμη, πρώτα κύριο Σμιθ. Πρώτα κύριο Σμιθ και μετά εσείς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ε, μπορούμε να κάνουμε <laughs> μια τελεγή εδώ μεταξύ Βρετανών. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε στα σχόλιά μου γιατί 100% ε, η ε, συμμαχία μας ε, λαμβάνει συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όσοι, προ... όσοι προωθούν τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς ε, ε, προσπαθούν να παρουσιάσουν ε, όσους είναι αντίθετους με τους γοναταφόμικρων ως ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν βάσει του συναισθήματος. Αυτό είναι προσβλητικό και δεν ε, ε, μιλάμε ε, εμείς ε, ε, με θεολογικούς όρους και με άσχημους όρους κατά των ανθρώπων οι οποίοι υποστηρίζουν τους γενετικά τρόπιμους οργανισμούς. Εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να τοποθετηθεί επί αυτής της πρότασης της Κομισιόν και πρέπει να τροφοδοτήσουμε με την γνωμοδότησή μας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εδώ διαφωνώ λοιπόν με τον συντάκτη ε, ε, ε, ε, φαίνεται σαν να υπάρχει μια αναγκαιότητα για να σταματήσει η τελμάτωση. Όμως αυτό είναι λάθος γιατί η πλειοψηφία των κρατών μελών και των πολιτών είναι κατά της καλλιέργειας των γαματόφων μικρών. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια, ε, ότι αυτή η πρόταση αποτελεί τελευταία προσπάθεια του λόμπι ε, των γαματαφόμικρων ε, να παρακάψουν όλα τα μέτρα προστασίας που έχουμε. Όλοι είμαστε στην νέα αγορά, αλλά εδώ προσποιούμαστε ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς κανόνες και να επιτρέψουμε στην επιμόλυνση να κάνει τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, εμείς απορρίπτουμε αυτή την πρόταση από την αρχή. Δεν θέλουμε εδώ να προσποιούμαστε ότι μία κακή πρόταση θα την κάνουμε καλύτερη. Αμέσως, από την αρχή πρέπει να την απορρίψουμε. Μάλιστα κύριε Σμίτ, Σα ευχαριστώ πολύ. Άσχορτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βλέπετε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, διαφορετικές νομικές απόψεις αλλά και συναισθήματα που προκύπτουν ε, Βάση αυτή τη συζήτηση. Ε, η γνωμοδότησή μα πρέπει να βασίζεται όμω σε δύο αρχές. Καταρχήν, οι αποφάσει ε, πρέπει να βασίζονται σε ε, αποδεικτικά επιστημονικά στοιχεία και δεύτερον πρέπει να σέβονται ε, την ελευθερία επιλογή και του παραγωγού και του καταναλωτή. Διάβασα τι προτάσεις του εισηγητή και πιστεύω ότι στι συγκεκριμένε συνθήκε είναι ρεαλιστικέ και αναλογικέ. Νομίζω ότι ήδη δίκαιο έχει που λέει ότι ο συνολικός κανονισμός ε, θα ε, πρέπει ε, να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται και αποφάσει και σε επίπεδο κρατών μέλου. Εγώ λοιπόν ε, θέλω να υποστηρίξω τι προτάσει του. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Κάπουλα Σάντος για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον μιλητή. Εγώ ζητώ συγγνώμη που δεν ε, συμμετείχα στη συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη που δεν συμμετείχα στην όλη συζήτηση, αλλά θα έπρεπε να ήμουν παρόν και στην Επιτροπή Αλία γιατί παρουσίαζα μια γνωμοδότηση. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ λεπτό και η δική μου πολιτική ομάδα έχει πολύ υπεύθυνη και σοφρόνα στάση στο εσωτερικό της δικής μας πολιτικής ομάδας μεταξύ βουλευτών από διάφορε επιτροπές προβαίνουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν ε, πιο κοινά συμπεράσματα. Θέλουμε να ε, εγγυθούμε τις νόμιμες ανησυχίες των πολιτών ε, σχετικά με όλα σου να κάνουμε με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και να δούμε σε ποιο σημείο ε, μπορούν να προστατευτούν ε, αποδεκτοί οι κανόνες ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Δεχόμαστε τη θέση που μόλις εξέφρασε ο συγητής ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και το θέμα της ελεύθερης επιλογής, αλλά φυσικά έχουμε και περιβαλλοντικές πτυχές που πρέπει να σκεφτούμε. Τώρα δεν θα τοποθετηθώ για κάθε μία από τις τροπολογίες, απλά μπορώ να σας πω ότι ε, η ομάδα των σοσιαλιστών ε, θα είναι διαθέσιμη για να καταλήξουμε σε έναν υπεύθυνο συμβιβασμό γύρω από ένα θέμα το ευαίσθητο, γιατί θεωρώ ότι μία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα είναι υπεύθυνη, θα συνεισφέρει έτσι ώστε αυτό το θέμα ε, να αντιμετωπιστεί και στην κοινή γνώμη με την υπευθυνότητα που του αξίζει και όχι με τον παραλογισμό που πολλές φορές γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λουίς. Κυρία Λούλινγκ. Συγγνώμη πρόεδρα που καθυστέρησα έπρεπε να πάω και σε άλλες δυο συνεδριάσεις. Ζήτησα το λόγο για να πω ε, πολύ γρήγορα ότι η κυβέρνηση της χώρας μου ε, ανήκει σε εκείνο το στρατόπεδο που δεν τους αρέσουν πολύ τα γενετικά τροποποιημένα γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Θα ήθελα να σας πω ότι στις αρχές δεκαετίας του 90 πήγα σε ένα σεμινάριο με την Επιτροπή Βιομηχανίας κοντά στη Washington όπου μας ε, έδειξαν και μας εξήγησαν πολλά πράγματα και μας και πήγα και σε ένα γεύμα όπου σερβιρίστηκαν μόνο προϊόντα, μη, ε, ε, προϊόντα γενετικά τροποποιημένα. Είμαι ακόμη ζωντανή, άρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να θεωρούμε τόσο πολύ επικίνδυνα τα προϊόντα αυτά. Συμφωνώ με άλλα λόγια γενικά με τη γενική γραμμή του εισηγητή. Μάλιστα, ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Ε, τώρα θα ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να πάρει το λόγο. Από την εκπρόσωπο τη Κομισιόν, μάλλον πάρει το λόγο, κυρία Αντρέ. Εδώ είστε μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την εργασία που έκανε ο εισηγητή σα. Γίνονται εδώ πέρα κάποιες προτάσεις βελτίωσης. Αυτό που θέλουμε να διευκρινίσουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται για τον περίφημο αυτό κατάλογο των other grounds, λυπή άλλοι λόγοι που θα μπορούσαν να επικαλεστούν τα κράτη-μέλη για να απαγορεύσουν την καλλιεργία γεντικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Ο κατάλογος αυτός θα δοθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύντομα και οι λόγοι αυτοί είναι λόγοι δεοντολογικοί, κοινωνικο-οικονομικοί, λόγοι περιβαλλοντικής πολιτικής με την ευρία έννοια του όρου και αυτό που είπε και ο συντάκτης της γνωμοδότησης, ο εισηγητής σας και στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε λίγο είναι ότι η ΕΦΣΑ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αξιολογεί την περιβαλλοντική και υγειονομική διάσταση, θεωρούμε ότι θα πρέπει η αξιολόγηση αυτή, ο έλεγχος αυτός να μείνει σε κοινοτικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που θα μπορούσαν ε, να επικαλεστούν ως λόγο τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έρθει ως επιπρόσθετος λόγος σε αυτά τα οποία κάνει η ΕΦΣΑ. Τώρα όσον αφορά τα μέτρα συνύπαρξης. 15 είναι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν εγκρίνει τέτοιους κανόνες συνύπαρξη 15 λοιπόν τα κράτη-μέλη που έχουν εφαρμόσει τους κανόνες αυτούς. Για τα λοιπά θεωρούμε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και με ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε ποια συνέχεια θα δοθεί στην έκθεση αυτή, καθώς επίσης και ποιες θα είναι τροπολογίες που θα κατατεθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Αντρέ να σας επιμιλήσω ότι η προθεσμία για την καταστροφή των είναι στις 9 Φεβρουαρίου, 15 Μαρτίου η ψηφοφορία. Και να δώσω το λόγο στον Τζόρτζ για να κλείσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους ε, που συνεισφέρατε στη συζήτηση. Πολλές δημιουργήθηκαν. Ίσως ε, να απαντήσω σε ένα-δύο, με τόσο ακούστηκαν. Είπατε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη, ε, κύριε Μποβέ, δεν θέλουν ε, την ε, πρόταση. Όμως εδώ, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, από το πιστεύει το Συμβούλιο, εμείς πρέπει να καταλήξουμε στη δική μας θέση. Θα τοποθετούμε ως Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, για θέματα εσωτερική αγορά. Ε, προσπαθήσαμε να ενδυναμώσουμε την νέα αγορά με τις τροπολογίες που κάνουμε, που υποβάλλουμε. Υπάρχει και συζήτηση για την ε, κοινή γνώμη. Νομίζω ότι ο κίνδυνος αυτής της συζήτησης ε, είναι εξή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν αρχίζουμε να λαμβάνουμε αποφάσει για την ασφαλεία των τροφίμων βάσει με όσων είναι δημοφιλή αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ε, πρέπει πάντοτε να βασιζόμαστε στις επιστημονικές αποδείξεις. Κάποιοι αναφέρθηκαν στο ότι υπάρχουν αποκλίνουσες επιστημονικές απόψεις. Η ακρόση που είχαμε πριν δύο-τρεις εβδομάδες, στην οποία προέδρευσα εγώ και η κυρία Λεπάς, ανέδειξε ότι να υπάρχουν αποκλίνουσες ε, επιστημονικές απόψεις αλλά όλες οι απόψεις έχουν ληφθεί υπόψη από την ΕΦΣΑ και κατά τη διαδικασία της έγκρισης ε, δόθηκαν και κατάλληλες απαντήσεις. Η ΕΦΣΑ δεν δέχτηκε όλες τις απόψεις, αλλά ορισμένες. Και αν υπάρχει διαφορά απόψεων, ε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι με τα πάντα. Το θέμα είναι τι απόφαση πήρε η ΕΦΣΑ. Ε, αναφέρεται ότι ε, ε, πρέπει να έχουμε κανόνες, συγκεκριμένως τον γνωρίζω αυτό. Υπήρξε και μία αναφορά στην πρόταση της Κομισιόν σε σχέση με τις χώρες. Όχι, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα κρατημέλη, μονόμενα κρατημέλη. Ο κύριος Σμιθ ανέφερε κάποιες ανησυχίες που είχε και είπε στο ότι πρέπει να έχουμε απευθείας απόρριψη. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με το ότι πιστεύει η κυβέρνηση της Σκοτίας που θέλει να υποστηρίξει ε, την προσέγγιση της, ε, του καταμερισμού των εξουσιών στην, ε, στις τοπικές κυβερνήσεις. Ε, άλλος, η κυρία Λούλινγκ είπε ότι ε, κάθε φορά που κάποιος ε, καταναλώνει ε, προϊόντα στην Ευρώπη δεν μπορεί να γνωρίζει σίγουρα αν έχουν χρησιμοποιηθεί γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Πολλές φορές πρέπει να το επισημαίνουμε αυτό στο κοινό Νομίζω ότι το αν η Ευρώπη έχει απόλυτο δίκιο πρέπει να το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ για το ότι δώσατε μεγαλύτερη προθεσμία για τις τροπολογίες, γιατί σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να καταλήξω σε συμβασμού, αλλά βέβαια θα βάλω το δυνατά μου για να διασφαλίσω ότι θα το πράξουμε. Ε, ευχαριστώ τον Τζόρτζ. Σημείο 6. Η Ευρώπη, πρώτο τουριστικό πολιτισμό στον κόσμο. Ένα νέο πλαίσιο πολιτική για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Η ο αντιπρόεδρο Νικολέσκο. Πρόκειται εδώ για μια πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Ε, ο αγροτουρισμός είναι μια πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα και ε, έτσι πρέπει να εγγυηθούμε την ανάπτυξή του μέσω στοχευμένων ε, μέτρων στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ μετά το 2013. Για το λόγο αυτό θα δώσω απευθείας το λόγο στον κύριο Νικονέσκου και χαιρετίζω την εκπρόσωπο της Κομισιόν, την κυρία Μπόρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόταση γνωμοδότηση έχει μεταφραστεί σε όλε τι γλώσσε και έχει διανεμηθεί. Έτσι λοιπόν ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Έχω λάβει και τις προτάσεις των συναδέλφων. Ε, εδώ ε, αναφερόμαστε στη στήριξη του αγροτουρισμού. Είναι κάτι σημαντικό στο πλαίσιο της πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό θέλουμε να διαφοροποιήσουμε την αγροτική οικονομία και επίσης ο αγροτουρισμός μας επιτρέπει ε, να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο της εγκατάλειψης των αγροτικών περιοχών από τον πληθυσμό. Ε, ο αγροτουρισμός είναι σημαντική δραστηριότητα για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των περιοχών και επίσης λαμβάνουμε υπόψη τη συνεισφορά του αγροτουρισμού για την ε, διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των εθήμων ε, των διάφορων περιφερειών. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις και αυτές θα παρουσιάσουμε στην ε, Επιτροπή Τουρισμού η οποία είναι η καθήλυν αρμόδια και χρειάζεται και χρηματοοικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ για το ζήτημα αυτό, όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος. Η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η 3η Φεβρουαρίου και αν έχετε προτάσει είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Τρει ε, Φεβρουαρίου, λίγη προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών, 28 Φεβρουαρίου, η ψηφοφορία. Α περάσουμε στη συζήτηση. Σέρζιο Γκουτιέρε, Έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Ουσιαστικά συμφωνούμε με τον κύριο Νικολέσκου, αλλά θέλω να παρουσιάσω και κάποιες περαιτέρω ιδέες, να ενισχύσω κάποια περαιτέρω ιδέα, γιατί θεωρούμε τον ε, τουρισμό στρατηγικό τομέα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να διαφοροποιήσουμε την οικονομία. Ένα είναι τομέα με τεράστια δυναμική και ε, ως ποσοστό ε, του ΕΠ ε, αλλά και ως ένα τομέα που συνεισφέρει άμεσα ή έμεσα στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να απευθύνουμε μια έκκληση για να έχουμε καλύτερες δημόσιες δράσεις από το συντονισμό αλλά και με τον να αναλάβουν ηγετικό ρόλο οι δημόσιες υπηρεσίες και να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Γιατί ο τουρισμός Εμ... Ε, θα μπορέσει να συνεισφέρει και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μα για πολλού λόγου. Καταρχήν για τη διαφοροποίηση τη οικονομία, γιατί θέτει νέε ευκαιρίε για του νέου και για τι γυναίκε πιο συγκεκριμένα. Γιατί ε, έχουμε συμπληρωματικέ δραστηριότητε ε, στι δραστηριότητε του πρωτογενού τομέα και μάλιστα στην περίπτωση του αγροτουρισμού ενισχύονται οι δραστηριότητε αυτέ. Επίση πρέπει να τονίσουμε ότι ο αγροτουρισμό και ο αγροτικό τουρισμό επιτρέπουν την οργάνωση των εργασιών εργασιών με νέε μορφέ που επιτρέπουν την ανάπτυξη τη κοινωνική οικονομία. Και αυτό μπορεί να έχει καλύτερη, ε, μεγαλύτερο αντίκτυπο στην απασχόληση. Ε, ο αγροτουρισμό ε, είναι ένα καθαρό τομέα και σε διαφοροποίηση με άλλων μοντέλων ευρωπαϊκού τουρισμού όπως ο τουρισμός στις ακτές επιτρέπει ε, ουσιαστικά καλύτερη ποιότητα τουρισμού και μπορεί να οδηγήσει και στην ανάπτυξη με περισσότερων θέσεων εργασία. Εμεί θα παρουσιάσουμε κάποιε τροπολογίε στην έκθεση Νικόλα Καταρχήν, ανταγωνιστικότητα του αγροτουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στοιχηματίσουμε για τον εξυγχρονισμό τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά και δύο κύριε ιδέε να βελτιωθεί το δίκτυο των μεταφορών στην Ήπεθρο, όχι μόνο από τη σκοπιά των υποδομών, αλλά και των δημοσίων υπηρεσιών. Και κυρίως είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την καινοτομία και δίνει εν ω ως ε, τομείς ανταγωνιστικότητας του αγροτουρισμού. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι τα περισσότερε θέσει εργασία ε, ε, σε αυτές τις επιχειρήσεις στην Ήπεθρο υλοποιούνται μέσω από πολύ μικρές επιχειρήσεις και όπω σα είπα απασχολούν ιδιαίτερα του νους και τι γυναίκε. και έτσι λοιπόν η δημιουργία μέσων που να βελτιώνουν τα προσόντα του προσωπικού μπορεί να οδηγήσει και στη δημιουργία και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και επίση θα πρέπει να αποτελεί ο αγροτουρισμός μέρος του κοινωνικού τουρισμού. Όταν ε, έχουμε έναν ε, τουρισμό που να απευθύνεται και στα άτομα περιορισμένης κινητικότητα, αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ε, σήμερα ε, στον αγροτουρισμό. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε ό,τι φορά την προσβασιμότητά του στα άτομα με ειδικές ανάγκες και αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να πληρούμε και κάποιους πολύ σημαντικούς κοινωνικούς στόχους. Ε, θέλουμε να στοιχηματίσουμε για την αριστεία. Έτσι λοιπόν πρέπει να εισαγάγουμε καλύτερη σχέση μεταξύ του αγροτουρισμού και του δικτύου Natura 2000 και να καθορίσουμε κριτήρια ομοιομορφίας στη στιγμή που θα καθορίζουμε σήματα ποιότητας ε, όπως ε, υπάρχουν σήμερα σε ορισμένους τομείς εκεί ε, για να δίνονται συγκεκριμένα σήματα, ε, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη ε, στους ξενώνες, εκεί πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια και πρέπει τον αγροτουρισμό να εντάξουμε με οριζόντιο τρόπο σε όλες ε, τις δράσεις που υποστηρίζουν τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια στρατηγική προτείνεται για τον τουρισμό στις ακτές να οργανώνει με οριζόντιο τρόπο όλα τα μέτρα που μπορούν να αναλάβουν από κοινού τα ευρωπαϊκά όργανα για να προωθήσουν και τον αγροτουρισμό. Δεν μπορούμε να πέσουμε στο λάθος να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική που θα θέτει ως κύριο άξονα ε, τη κοινοτικής δράση, ε, μόνο τον τουρισμό στις πόλεις ή τον τουρισμό στις ακτές. Και να παρουσιάσω και μια ιδέα, να ενισχύσω μια ιδέα που ανέφερε ο κ. Νικολέσκου. Είναι αλήθεια, όπως ε, λέει η Κομισιόν. Ε, τονίζει τη σημασία που είχε το έκτυπε κατά την ανάπτυξη του αγροτουρισμού πρέπει να έχει και το έκτυπε την κατάλληλη πρικοδότηση, δηλαδή να μην ε, ε, μιλάμε μόνο για το δεύτερο πυλώνα, αλλά κάτι πιο σημαντικό. Όλοι γνωρίζουμε ε, ότι οι πολίτες δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο, να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στην κυρία Κριστίνα Μπόρος. Uh, uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα η Επιτροπή θα ήθελα να ευχαριστήσει την Επιτροπή σας που συζήτησε το θέμα αυτό και αναγνώρισε τη σημασία του τουρισμού. Και εμείς ενδιαφερόμαστε προφανώς τον τουρισμό, με για τον τουρισμό, για, ιδιαίτερα για τον αγροτουρισμό, αναγνωρίζουμε και αναγνωρίσαμε, αναγνωρίζουμε τη σημασία του κλάδου αυτού στην οικονομία και βλέπουμε ότι ο αγροτουρισμός μπορεί να αλλάξει και να διαφοροποιήσει αν θέλετε ολόκληρες περιοχές της υπαίθρου μας. Από την άλλη μεριά είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά όλοι μας και τις, δια... τις ιδιαιτερότητές μας. Για να προωθήσουμε τον τουρισμό λοιπόν και να κάνουμε όλα αυτά, μια ιδέα θα ήταν να προωθήσουμε καινοτόμε πρωτοβουλίες όπως αναφέρει και ο εισηγητής, να βοηθήσουμε τις μικροεπιχειρήσεις που είναι παρούσες στις, ε, σε κάποιες περιοχές της υπαίθρου, να τις βοηθήσουμε λοιπόν να συμμετάσχουν στην αλυσίδα ε, προσφοράς ε, την ψηφιακή. Ξέρουμε ότι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή οι μικρές επιχειρήσεις στην Ήπεθρο δεν έχουν, έχουν κάποια προβλήματα ε, στο να παράσχουν τα προϊόντα του ή να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε ε, διαφορετικά τόπους άρα αυτό θα μπορούσε να τους βοηθήσει επίσης θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την κινητικότητα ιδιαίτερα σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές και μειονεκτικές περιοχές γιατί και αυτό θα βοηθούσε την όλη υπόθεση κάτι τι άλλο Για το καλύψω, όπως λέμε στην ε, πρόταση, ε, πρόκειται πρώτα-πρώτα για μια πρωτοβουλία που έχει σε στόχο να αντιτεθεί στην εποχιακότητα, αν θέλετε. Να βοηθήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες ε, τους ηλικιωμένους, τους στοχότερους και τα λοιπά ή τους, ε, ε, τα άτομα με αναπηρίες να ε, απολαύσουν τον τουρισμό άσχετα από την εποχή αν θέλετε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης υπάρχει και μια άλλη πρωτοβουλία για την ε, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς υπάρχει άλλη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας, υπάρχει πρωτοβουλία σχετικά με τις συνέργειες και ιδιαίτερα με τη, συνέ, ε, με τη συνέργεια με το Natura 2000 ελπίζουμε πραγματικά όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να προωθηθούν και να υποστηριχθούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα και ε, νομίζω ότι θα συνεργαστούμε καλά στο μέλλον. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Νικολέσκου, δεν θέλει να παρέμβει και να Σα υπενθυμίσουμε ότι θα ξανασυναντήσουμε την επόμενη Δευτέρα στι 7 Φεβρουαρίου στι 3. Σα ευχαριστώ όλου Λήξη τη συνεδρία σας.